Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε τώρα με την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής ΠΕΜ. Αρχικά, η έγκριση της τη διάθεσης, σε περίπτωση λοιπόν που δεν υπάρχουν σχόλια, θεωρείται ότι εγκρίνεται. Στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών της 3 η Σεπτεμβρίου και της 27ης Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχουν σχόλια, οπότε εγκρίνονται. Τέταρτον, ε, ανακοινώση του Προέδρου. Στην συνάντηση τη 8η Νοεμβρίου, οι συντονιστέ αποφάσισαν να υποβάλουν ένα προφορικό ερώτημα, το οποίο θα ακολουθηθεί από ψήφισμα σχετικά με το ρόλο των γυναικών στην αποτροπή τη ακρεοποίηση ε, και να δοθεί στην ομάδα του ΕΛΚ. Το έργο αυτό θα περιοριστεί σε επίπεδο επιτροπή. Το σημείο 5 τώρα της ημερήσιας διάταξης αφορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Mm. Ε, ε, ε, Σημείο 5 λοιπόν τη ημερήσια διάταξη, η θέσπιση του προγράμματο για τα δικαιώματα και τη αξία. Συντάκτρια τη ομοδότηση ήταν η κυρία Σύρπα Πιετικάινεν. Και τώρα θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Τροπολογία 54 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ, Ε, Άκουσα στην αρχή 55 και ήταν η 54. Μπορούμε να ξανακάνουμε την ψηφοφορία παρακαλώ γιατί μπερδεύτηκα με τα νούμερα. Yes, we will start. Ναι, θα αρχίσουμε και πάλι από την αρχή. Τροπολογία 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 66 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 58 όχι, πηγαίνουμε στην συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστικές 7 και 8 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 72. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 75 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 και 83 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 και 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 και 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά 12, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 110 και 11 υπέρ κατά αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε εδώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 112 υπέρ Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Είναι δυνατό, απαντάει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 112 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία Α, όχι, πάμε στην συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, δι, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά εγκρίνεται 28 υπέρ πίπτη οπότε πάμε στην συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 50 τοπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 51 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα ψηφίζουμε επί του συνόλου του κειμένου όπως έχει τροποποιηθεί άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Σύρπα Πιετικάιν και όλους τους σκιώδεις. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλες ψηφοφορίες στην ημερήσια διάταξη. Οπότε περνάμε στο σημείο 6, την αποστολή στην Αυστρία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και σχόλια, τότε θεωρείται ότι η έκθεση εγκρίνεται. Ωραία. Οπότε περνάμε στο σημείο 7 το οποίο αφορά ε, την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τους τριμερείς διαλόγους για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ένα λεπτάκι όμως να αδειάσει η αίθουσα. Mm. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Νιέσκα Κοσλόφσκα Ράγεβιτς που είναι η συγγήτρια για την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας όσον αφορά την ισορροπία αυτή μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω πολωνικά αν μου επιτρέπετε, οπότε βάλτε τα ακουστικά σας για να με καταλάβετε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πριν να αρχίσω, πρέπει να σας ενημερώσω για αυτό το πακέτο, αλλά να εκφράσω και την απογοήτευσή μου για τη συμπεριφορά που είχαμε εδώ Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας που κάναμε πριν από λίγο για την ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές, έχουμε δικαίωμα όλοι να έχουμε διαφορετικές απόψεις και εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε διαφορετικές απόψεις. Ετοιμάσαμε κάποιες τροπολογίες και οι άλλοι μας κοροϊδεύαν γι' αυτό. Κάνανε σχόλια εκτός μικροφώνου, κάπως προσβλητικά, εμείς τα ακούσαμε όμως αυτά. Λοιπόν, αυτή η συμπεριφορά με απογοήτευσε πολύ, γιατί η δημοκρατία υπάρχει αν δεν υπήρχε δεν θα είχαμε γνωμοδοτήσει. Λοιπόν, από τις ψηφοφορίες εξαρτάται πώς θα καταλήξει μια έκθεση. Εδώ η ομάδα που είχε τις περισσότερες ψήφους βέβαια κέρδισε. Πάντως η δικιά μας άποψη, πέρα από την μειοψηφούς άποψη, δεν θα μπορέσει να ενσωματωθεί αλλιώς στην έκθεση. Τώρα, έρχομαι στους τριμερείς διαλόγους. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ θετική. Παρόλο που στην αρχή οι θέσεις ήταν ε, αρκετά διαφορετικές μεταξύ μας, η θέση του Συμβουλίου, για παράδειγμα, είναι πολύ διαφορετική από εκείνη του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο ήθελε τέσσερις μήνες να έχει ατομικό δικαίωμα σε γονική άδεια η μητέρα ή ο πατέρας. Καταλήξαμε σε ένα 78% στο τέλος και είχαμε και 10 μέρες ε, ελοχίας πληρωμένη βέβαια και όλες αυτές οι άδειε θα έπρεπε να είναι ευέλικτες, δηλαδή να μπορεί κανείς να επωφεληθεί από αυτές τις μέρες μέχρι να κλείσει τα 10 χρόνια το παιδί. Είδαμε στην αρχή ότι η θέση του Συμβουλίου ήταν εντελώς διαφορετική από τη δική μας. Λέγανε ότι θέλαν 1,5 μήνο, μήνα πληρωμένη άδεια με αποδοχές. Αυτό ήταν το επίπεδο των χωρών μελών. 10 μέρες για τον πατέρα. Και δεν θέλανε τίποτα για φροντίδα κλπ. Τελικά το δέχτηκαν, παρόλο που πολλές χώρες ήταν κατά. Και βέβαια δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε για πληρωμή. Οι θέσεις μας λοιπόν ήταν πάρα πολύ διαφορετικές στην αρχή. Σιγά σιγά περιμέναμε ότι θα προσεγγίσουν οι θέσεις μας. Τελικά όμως έγινε το αντίθετο. Αντί να προσεγγίσουν οι θέσεις μας, απόκλειναν ακόμα περισσότερο. Υπήρξε μια συνάντηση Κορεπέρ όπου ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη να επιβεβαιώσουν τις θέσεις τους. Οι αλλαγές δεν οδήγησαν σε τίποτα όμως. Το μόνο σημείο που πετύχαμε κάποιο αποτέλεσμα, γιατί βρέθηκαν πιο κοντά στις θέσεις του Κοινοβουλίου, είναι στο θέμα ακριβώς της ε, πατρικής ε, άδειας. Δύο εβδομάδες με αποδοχές. Θέλανε η πληρωμή να γίνεται σε επίπεδο αναρωτικής. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το δεχτούμε, γιατί, εν πάση το επίπεδο αυτό είναι αρκετά ψηλό. Τώρα όμως έχουμε και άλλα προβλήματα, ακόμα και σε αυτό, γιατί το Συμβούλιο απέσυρε κάποιες από τις υποχωρήσεις που είχε κάνει προηγούμενα και στην τελευταία συνάντηση μας ζήτησε να ξαναδούμε τις θέσεις μας. Εμείς είπαμε ότι αυτές είναι. Έχουμε τις λεπτομέρειες από την διαπραγμάτευση και αν δεν υπάρξει κάποια προοπτική συμφωνίας, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Η γονική άδεια πάντως είναι το πιο βασικό για τις μητέρες και τους πατεράδες και να πληρώνεται βέβαια σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Εμεί είπαμε στο Συμβούλιο ότι πρέπει να το ξανακοιτάξει, γιατί πρέπει να υπάρχουν ε, διαπραγματεύσεις. Το θέμα δεν είναι να καθόμαστε να συζητάμε τις λεπτομέρειες για τη ρήτρα, πασαρέλα και τέτοια. Πρώτα πρέπει να έχουμε τα βασικά, να έχουμε συμφωνήσει πάνω στα βασικά. Οπότε αισιόδοξη δεν είμαι. Περνάει και ο χρόνος, φαίνεται να είμαστε σε αδιέξοδο. Τελειώνει και η Προεδρία αυτή. Αν το Δεκέμβριο δεν έχουμε ολοκληρώσει, θα έχουμε περάσει στην επόμενη Προεδρία και δεν ξέρω πόσου τριμερεί διαλόγου θα προλάβουμε να κάνουμε τότε, δύο το πολύ. Και με τι αποτελέσματα ποιο ξέρει. Θα προτιμούσα λοιπόν το Κοινοβούλιο να ήταν λιγότερα φιλόδοξο και να συμφωνήσει με περισσότερα για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, γιατί έτσι όπως πάμε τώρα δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Η οδηγία για τους γονείς δεν επιβάλλει τίποτα, κάνει μόνο συστάσεις. Και σε κάποιες χώρες δεν πληρώνεται καθόλου η γονική άδεια και δεν υπάρχει καθόλου άδεια για τον πατέρα. Νομίζω ότι έτσι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε, να κατεβάσουμε κάπως τις απαιτήσει μας. Ξέρω ότι υπάρχουν ομάδες που είναι εντελώς κατά τέτοιων ε, υποχωρήσεων και δεν θέλουν να συμφωνήσουμε με τίποτα. Να δεχτούμε δηλαδή αυτά που προσφέρει το Συμβούλιο. Θέλουν να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσει από την αρχή για όλα. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Πέρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, πριν μπούμε σε οτιδήποτε άλλο, θέλω να αναφερθώ λίγο στο θέμα της μετάφρασης αυτού του φακέλου. Την προηγούμενη εβδομάδα τι συνέβη. Στην έκθεση που αναφέρεται σε αυτούς που φροντίζουν άτομα που έχουν ανάγκη και εκεί που αναφερόμασταν στη γονική άδεια, στα ισπανικά μερικές φορές μεταφράζεται σαν ε, άδεια διακοπές σαν να πρόκειται για διακοπές. Και εμένα με απασχολεί πολύ αυτό, γιατί οποιοδήποτε πολίτη στην Ισπανία πάρει την έκθεση αυτή και εκεί που μιλάμε για τη γονική άδεια αναφέρεται στα ισπανικά ότι πρόκειται για διακοπές, ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι διαφορετικό, έτσι. Δεν έχει καμιά σχέση με τη φροντίδα που προσφέρουν τα άτομα αυτά στους δικούς τους. Ας κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια παρακαλώ. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και με άλλες γλώσσες, μου εξήγησαν ότι η λέξη στα αγγλικά leave μπορεί να σημαίνει και το ένα και το άλλο. Αλλά να προσέχουμε πολύ τη μετάφραση, τη διερμηνία, γιατί καταλαβαίνετε είναι εντελώς διαφορετικό να μιλάμε για διακοπές και εντελώς διαφορετικό να μιλάμε για άδεια προκειμένου να φροντίσει κάποιο τους δικούς του. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν ε, μεταφέραμε το μήνυμα στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω εκείνες να το μεταφέρουν ε, στις υπηρεσίες μετάφρασης. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα που ήθελα να πω. Δεύτερον, όσον αφορά τώρα την οδηγία αυτή για την ισορροπία επαγγελματική και προσωπικής ζωής. Η πρόταση αυτή οδηγίας, καταρχήν, έχει ως συνέπεια να μπλοκάρει άλλη οδηγία που για χρόνια ζητούσαμε. Εκείνη για την υγεία των γυναικών στην εργασία και για τις άδειες μητρότητας. Τι θέλω να πω, ότι μέρος της κατάστασης στην οποία εδώ και χρόνια βρισκόμαστε, επειδή εδώ και καιρό θέλουμε μια λύση για να επιτευχθεί ακριβώ αυτή η ισορροπία επαγγελματικής ε, και προσωπικής ζωής. Όμως το αποτέλεσμα ήταν ότι αποσύρθηκε αυτή η πρόταση. Άντε πάλι να το εξηγούμε αυτό στον κόσμο. Λες και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ισορροπία. Ε, δεν το κάνουμε. Περιμέναμε λοιπόν πάνω από ένα χρόνο, δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν, ώστε η Ευρωπαϊκή, η Επιτροπή να έρθει με την νέα πρόταση. Έρχεται λοιπόν με ένα πλαίσιο κοινωνικού πυλώνα, όπως το ονομάσαμε, όπου ζητούμε να συμπεριληφθούν διάφορα νομοθετικά θέματα και το μόνο καθαρά νομοθετικό είναι ακριβώς αυτό. Δεν βλέπουμε να υπάρχει δηλαδή δέσμευση να προχωρήσουμε πράγματι για τον κοινωνικό πυλώνα. Παρ' όλα αυτά είναι ευπρόσδεκτη η πρόταση. Όμως, τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό που δεν μπορεί να κάνει είναι να παραιτηθεί από τις βασικές αρχές της οδηγίας. Και γι' αυτό είναι οδηγία γιατί είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί. Και άκουσα τι είπε εκπρόσωπος του ΕΛΚ που λέει πόσο δύσκολες είναι οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ναι, αλλά αν το Κοινοβούλιο ήδη παρετηθεί από τις πολιτικές του θέσεις, τις οποίες συμφώνησε και με τις οποίες συμφωνούν όλοι, τότε τι κάνουμε, δεν φέρουμε σε πέρα στο ρόλο μας στις διαπραγματεύσεις του Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε στις θέσεις μας. Και έτσι να ξέρουν όλοι τι υποστηρίζουμε. Αν τώρα συγχρόνως ο καθένας από εμά μπορεί να πείσει τις εθνικές του κυβερνήσεις να τροποποιήσουν τις θέσεις του Συμβούλιο, τόσο το καλύτερο. Αυτό είναι το σημαντικό. Επιμένω πάντως, στο Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μας, οι Ευρωβουλευτές που έχουμε την ευθύνη να φέρουμε σε πέρα σημαντικές διαπραγματεύσεις, πρέπει να συνεχίσουμε και να επιμείνουμε στη θέση που υιοθετήσαμε και η οποία αντικατοπτρίζει και την πολιτική βούληση τη δικιά μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα η κυρία Μπιόρκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. να συμφωνήσω με τα όσα ελέγχθησαν και με τα όσα είπε ο εισηγητής. Η άδεια του 1,5 μήνα είναι μόνο για αγωνικές άδειε δηλαδή που θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Εγώ θα ενθάρρυνα τον εισηγητή να μην αποδεχθεί αυτές τις ε, σκαιές προτάσεις του Συμβουλίου. Πρέπει να έχουμε μια θέση από τις οποίες να μπορούμε να δουλέψουμε. Η κυρία Ζεμπόσκα. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με την Αγνιέσκα. όταν λέει ότι πρέπει να είναι εύλογα τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η Γκαρθία Πέρεθ και άλλοι εδώ αναφέρθηκαν στην ε, προστασία της υγείας των γυναικών και τις σχετικές διατάξεις σχετικά με τις γυναίκες ε, που έχουν παιδιά και τα θυλάζουν και τα λοιπά ακούω σχετικά με το υπερβολικό επίπεδο της φιλοδοξίας μας. Εδώ φτάνουμε στο τέλος της εντολής μας και η σχετική οδηγία νομίζω ότι ε, θα πάρει το δρόμο της αντίστοιχα. Ε, το θέμα είναι ότι το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει σε μια κατάσταση, σε ένα καθεστώς καλύτερο από το υφιστάμενο ίσως να έχουμε ένα βήμα πιο μικρό από αυτό που επιθυμούσαμε, αλλά ανάλογα με τα αποτελέσματα των εκλογών, η εναρμόνιση των υποχρεώσεων της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής θα μπορούσε να δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο ανάλογα με τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν. Αναφέρομαι και στην κυρία Γαρθία Πέρεθ, αρκετές διατάξεις αναφέρουν τη μητρική άδεια με διάφορες ονοματολογίες. Αν θέλετε να βρούμε μια καλύτερη ορολογία σχετικά με αυτούς που φροντίζουν παιδιά, ίσως να μας απελευθέρουν λίγο από το θέμα της ορολογίας της άδειας σχετικά, εν πάση περιπτώσει, με τους ανθρώπους αυτούς που έχουν αφιερώσει την προσοχή τους στα παιδιά. Εάν η Αγνίασκα θα μπορούσε να βρει μια άλλη λέξη, έναν άλλο όρο, θα μπορούσε αυτό να είναι ένα χρήσιμο βήμα προς τα εμπρός, γιατί τότε ίσως θα μπορούσαν θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να σεβόμαστε τις υποχρεώσεις των γονέων ως προς τα παιδιά σου. Σας ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Εξ τώρα της κυρίας Αρένα η οποία διαπραγματεύεται, μάλλον συμμετέχει στην τριμερή, στον τριμερή διάλογο. Η κυρία Αρένα δεν μπορεί να είναι μαζί μας και ζητάει συγγνώμη. Είναι μέλος της ΣΕΜΠΛ. Ζητάει λοιπόν συγγνώμη που δεν μπόρεσε να παραστεί στην συνεδρίασή μας, όμως με ενημέρωσε σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και θα ήθελα να σας διαβιβάσω την θέση της, την οποία εγώ προσωπικά υποστηρίζω. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμερούς διαλόγου 19 Νοεμβρίου το Συμβούλιο παρουσίασε την τελευταία του θέση, την τελευταία του εντολή η οποία όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί βήμα προς τα εμπρός, πρόοδος. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξηγήσαμε στο Συμβούλιο ότι δεν θα μπορέσει να, συνεχίσει, να συνεχιστεί αυτή η διαπραγμάτευση εφόσον επιμείνει το Συμβούλιο στη θέση του. Η κυρία Αρένα και εγώ θα θέλαμε να ζητήσουμε από τους συναδέλφους της Επιτροπής και όχι μόνο αυτής της Επιτροπής να ασκήσουν μια, την πίεση εν πάση που μπορούν προς τα κράτη-μέλη προφανώς κάναμε κάποιες παραχωρήσεις αλλά δεν λάβαμε επαρκείς αντισταθμίσεις. Και όπως εξήγησε η κυρία Αρένα, αποφασίσαμε να διακόψουμε τον τριμερή διάλογο. Υπάρχει ακόμα κάποιος χρόνος πριν από τον επόμενο τριμερή 3 Δεκεμβρίου και επομένως την ε, υποστήριξή σας να ασκηθεί μια πίεση στις κυβερνήσεις των κρατών μελών για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα αυτό που να μπορούμε να υποβάλουμε στους πολίτες. Διότι πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα που άπτεται των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Τώρα, ε, ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία στην Ανιέσκα για την υπόλοιπη διαπραγματεύση. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά είναι σημαντικό να φτάσουμε, όπως έλεγα, σε ένα θετικό το αποτέλεσμα. Τώρα, κλείσαμε με αυτό το ζήτημα. Έχουμε και το μέσο διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης. Ελεονόρα Φορένζα έχει αργήσει. Άρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Θα πάμε στο επόμενο σημείο. Γενικός Προϋπολογισμός. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μπιόρκ είναι η συγητής. Η κυρία Μπιόρκ, συγγνώμη στην οποία θα δώσω τώρα το λόγο παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφός μου, κυρία Ρεφερέντσα, έχει αργήσει λιγάκι, οπότε θα μπορούσα πρώτα να ε, παρουσιάσω τα δικά μου δύο θέματα. Αρχικά αφορά την απαλλαγή ε, για τον τίτλο 3 ε, με την Επιτροπή και τις ε, υπηρεσίες. Ε, όπως βλέπετε, έχω συντάξει μια σύντομη γνωμοδότηση. Αυτό το οποίο όμως θα ήθελα να τονίσω είναι, όσον αφορά την απειλαγή είναι ότι η Επιτροπή μας θα ήθελε να διασφαλιστεί το ζήτημα των επενδύσεων για την ισότητα των φύλων και γι' αυτό το λίγο λόγο καλό την Επιτροπή BADS να επικεντρωθεί στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Δάφνη, τα ε, δικαιώματα της αναπαραγωγικής υγείας, ε, ε, αυτό όσον αφορά τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση και πιστεύω λοιπόν ότι όταν εξετάζουμε την απαλλαγή ε, θα πρέπει να ε, δούμε το πώς δαπανώνται οι προπολογισμοί τόσο όσον αφορά συγκεκριμένες ε, επενδύσεις αλλά και όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Και επίσης αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να μιλήσω και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων. Και εδώ προτείνω απαλλαγή ε, και έχουμε ε, κάποια σχόλια. Το Ινστιτούτο αυτό έχει ακολουθήσει τους ε, κανονισμούς και τονίζω το πόσο σημαντικό είναι το να έχουμε το συγκεκριμένο Ινστιτούτο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη δουλειά μας και έχουμε μια πολύ σημαντική έκθεση σχετικά με το trafficking ε, και, την, ε, και το ζήτημα της διάστασης του φύλου σε αυτό το θέμα και επίσης αναφέρθηκα και στην έκθεση σχετικά με την ε, σεξουαλική παρενόχληση ε, το οποίο επίσης είναι μια έκθεση που έχει δημοσιευθεί από, την, ε, από το συγκεκριμένο Ινστιτούτο ε, και έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα και έχουν προσπαθήσει να αναφερθούν στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Γι' αυτό το λόγο και εδώ προτείνω να υπάρξει απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φίλων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βιόρκ. κυρία Μετέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Μπιόρκ. Ως σκιώδης του ΕΛΚ ε, συμφωνώ με την εισηγήτρια για την εισαγωγή των δικαιωμάτων ε, των γυναικών ε, και των αρχών ισότητας στον γενικό προϋπολογισμό, όπως προβλέπει και ο Γενικός Κανονισμός, υποστηρίζω και την γραμμή για την ισότητα και τα δικαιώματα των πολιτών για το 14-20, όπως και εκείνη που προβλέπεται για το πρόγραμμα Δάφνη, προκειμένου να καταδειχθεί η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της ε, βίας κατά των γυναικών. Εμείς πάντοτε εργαζόμαστε επ' αυτού και το πιο έντονο σινιάλο που μπορούμε να διαβάσουμε στους πολίτες μας είναι ακριβώς η υποστήριξή μας προς τα προγράμματα αυτά. Τα οποία αφορούν άμεσα ή στην καθημερινότητά τους και είναι μία από τις βασικότερες στοχεύσεις μας. Εγώ, όπως πάντα, είμαι ανοιχτή σε έναν επικοδομητικό διάλογο και σε τροπολογίες εξίσου επικοδομητικές για να βελτιωθεί η θέση μας χωρίς να επιβαρύνονται αυτά τα προγράμματα από τον προϋπολογισμό. Για την ε, απαλλαγή, επιτρέψτε μου να πω στην κυρία Μπιόρκ ότι και εδώ είχαμε μια ισορροπημένη δουλειά και όχι υπερβολικά ιδεολογική. Αυτοί που με γνωρίζουν ε, ξέρουν ότι εγώ δεν τοποθετώ τις, ε, σημα... τις πολιτικές σημαίες, τις κομματικές σημαίες μπροστά από τόσο σημαντικά ζητήματα. και μπροστά στις εξελίξεις των επομένων ετών πρέπει να ξεπεράσουμε ίσως κάποιες κομματικές περιχαρακώσεις. Μιλούμε εδώ για το κοινό μας συμφέρον. Πρόκειται για ένα θεσμό θεμελιώδους σημασίας για όλους εμάς εδώ στο Κοινοβούλιο και που έχει και θετικό αντίκτυπο στην επικράτεια. Και το ελεγκτικό συνέδριο μάλιστα ε, συγχαίρει τον οργανισμό αυτόν και επομένως απόλυτη υποστήριξη ως αυτό από πλευράς μας. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ματέρα. Η κυρία Σπιτσέρνα. Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ να συγχαρώ την ε, κυρία Μπιόρκ για την δουλειά αυτή, για τις προτάσεις προς τις οποίες συμφωνώ απολύτως. Ήθελα να υπογραμμίσω ότι η εκτέλεση του προϋπολισμού για την ισότητα των φύλων δεν μπορεί ε, να μας ικανοποιεί πλήρως, ιδιαίτερα καθότι στο πρόγραμμα ισότητα ε, δεν υπάρχουν οι συγκεκριμένες στοχεύσεις των επιμέρους αντικειμένων το οποίο καθιστά και την εξπόστα αξιολόγηση λίγο πιο περίπλοκη. Η προσπάθεια του Κοινοβουλίου εδώ και χρόνια να υπάρχει συγκεκριμένη πίστοση πρόβλεψη του προεπολισμού ή το Δάφνη, προς αυτό αποσκοπούσαν. Να υπάρχει καλύτερη σαφήνεια σχετικά με τα αντικείμενα που επιδιώκουμε. Δεν είναι μόνο θέμα αρχής δηλαδή. Αλλά και πρακτικών διευθετήσεων, λειτουργικότητος. Όπω η εξπόστα αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης των κονδυλίων αυτών. Επομένως, είναι σημαντικό, θεωρώ, σε όλα τα κεφάλαια του προπολογισμού, και ούτως ή άλλω έχουμε ήδη ανταλλάξει ε, θέσεις και ιδέες και προτάσεις επ' αυτού, να έχουμε μια οριζόντια, ε, θα λέει κανεί προσέγγιση και αυτό θα πρέπει να το επιτηρήσουμε και με την ε, συλλογή δεδομένων που θα είναι διακριτά ως προς το φύλλο. Και ε, για το επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως και εκ μέρους του, της σκιώδους εισηγήτριας των SND που δεν μπορούσε εδώ να είναι σήμερα η Γκαμπριέλα Τζοάννα ευχαριστεί την εισηγήτρια για τις προσπάθειές της. Συμφωνεί με το σχέδιο αυτογνωμοδότησης, ήθελε να υπογραμμέσει την σημασία του ΛΕΓ και την πολύτιμη έρευνά του για την Επιτροπή ΦΑΜ, για την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, τις ανισότητες τις εισοδηματικές και πολύ χαιρόμαστε ότι που θα επικαιροποιούνται ετησίως οι δείκτες από το 19 και μετά. Οι δείκτες για την ισότητα. Επίσης ο οργανισμός για τα εσωτερικά θέματα λαμβάνει, βλέπουμε υπόψη του επαρκώς τα θέματα ε, και στον πεδίο της μετανάστευσης και του ασύλου είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε καλύτερα και με τι υπόλοιπε επιτροπέ του Κοινοβουλίου, ώστε η διάσταση αυτή να ενσωματώνεται καλύτερα σε όλες τις πολιτικές και δράσει. Το ΛΕΓΚΕ θα έπρεπε να έχει την ε, ανάθεση, την εντολή, στα πλαίσια τη ε, σύμβαση Κωνσταντινούπολη ε, να παρακολουθεί τα θέματα τη ισότητα των φύλων. Γνωρίζουμε βεβαίω τον διαρκή κίνδυνο και τη διαρκή απειλή τη περικοπής των πόρων, ε, το οποίο θα έχει αντίκτυπο επί του Λέγκε και στο πεδίο των ανθρωπίνων πόρων για να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την έρευνά του για την ισότητα των φύλων, το οποίο είναι απαράδεκτο και θα θέλαμε να ζητήσουμε πρόσθετη χρηματική στήριξη προς τον οργανισμό για να αυξηθεί το προσωπικό του, ώστε να είναι ακόμη πιο αποτελεσματική η δουλειά που κάνει το κέντρο έρευνας, το οποίο θα μας επιτρέψει να βοηθήσουμε τους ενδιαφερόμενους φορείς ε, και την σημαντική δουλειά που κάνουν. Η Γκαμπριέλα θα υποβάλει κάποιες τροπολογίες επί των θεματικών αυτών που ανέφερα και βεβαίως με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση θα συνεργαστεί με την εισηγήτρια και όποιον άλλο συνάδελφο ενδιαφέρεται για το θέμα. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βιόρκα. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Ναι, όντως θα έχουμε μια πολύ καλή ε, έκθεση και, για τον, ε, και όσον αφορά την απαλλαγή των προπολογισμού, όσον αφορά και την ΑΕΚ και όλοι εμείς που είμαστε ε, φεμινιστές και φεμινίστριες ε, θα πραγματικά απαιτούμε προϋπολογισμούς, ε, απαιτούμε οι ε, δραστηριότητες μας να έχουν τους απαραίτητους πόρους ε, και θεωρώ ότι μόνο όταν αγωνιζόμαστε για την ισότητα και ασχολούμαστε με αυτά τα σημαντικά ζητήματα του προϋπολογισμού, τότε μονάχα μπορούμε να επιτύχουμε κάτι. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τις τροπολογίες σας που συνεισφέρουν σε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Στι στις 30 Νοεμβρίου μπορείτε μέχρι τότε να ε, υποβάλλετε τροπολογίες τόσο όσον αφορά τον, από, την απαλλαγή όσο και τον γενικό προϋπολογισμό ε, της Ένωσης αλλά και την υπηρεσία ΕΓΕ Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περιμένουμε να έρθει η κυρία Ελεονόρα Φορέντσα. οι συνάδελφοί μου με ενημέρωσαν ότι θα είναι εδώ στις 10 και μισή. Συγγνώμη για αυτό, επαφείτε στην Προεδρία και τα μέλη να αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουμε. Θα σταματήσουμε λοιπόν τώρα για 10 λεπτάκια και θα περιμένουμε μέχρι ότου έρθει η κυρία Ελεονόρα Φορέντσα. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν με την ε, ε, συνεδρίασή μας ε, στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης σχετικά με το Εργαλείο Διεθνούς Συνεργασίας. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ελεονόρα Φορέντσα, συζήτηση περί των τροπολογιών και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην συγγήτρια. Κυρία Φορέντσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την ε, αναμονή και ζητώ συγγνώμη. Να ευχαριστήσω και τους ε, σκιώδεις ε, για την συνεισφορά τους στην διάταξη αυτή γιατί το να εργάζεται κανείς επί κανονισμού γνωρίζετε, καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη δουλειά. Νομίζω ότι μέσω των διαφορών τροπολογιών καταφέραμε να συνεισφέρουμε σημαντικά ως προς την εντολή της Επιτροπής μας. Αρχικά ο κανονισμός αυτός δεν είχε ιδιαίτερες ε, αποχρώσεις ως προς την ισότητα του φύλου. Νομίζω ότι ουσιαστικά βελτιώσαμε το κείμενο πρώτης ψήφου παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή ΦΑΜ έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα, υπάρχουν ζητήματα επί των οποίων είναι επίγον και είναι απαραίτητο να διαβιβάσουμε ένα μήνυμα μεταξύ των οποίων τα θέματα μετανάστευση Συζητούμε για τη συνεργασία με γειτονικέ χώρες ή στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων για την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Νομίζω ότι στο Κοινοβούλιο αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι οι θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ελπίζουμε λοιπόν να γίνει μια σημαντική προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή και να διαβαστεί αυτό το σημαντικό μήνυμα. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much, Ευχαριστούμε πολύ κυρία Φορέντσα. Παρακαλώ. Κύριε Χανιβό. Μιλάω εκ μέρου τη κυρία Μόντι, που είναι σκιώδη και πρέπει να είναι στην Επιτροπή Προπολογισμών στην ψηφοφορία. Σε τα συγγνώμη που δεν είναι εδώ. Και ο σκιώδη από του σοσιαλιστέ, η Κλέρ καλωσορίζει την δέσμευση του Κοινοβουλίου υπέρ της ισότητας και υπέρ της στήριξης των γυναικών και των κοριτσιών, αλλά και υπέρ της κοινότητας LGB. Πρέπει να ξέρουμε ότι δυστυχώς υπάρχει κάποιο πιστοχώρηση στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών και στα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα, αλλά αυτό το λέμε και αυτό είναι πολύ θετικό. Επίσης, πρέπει να προχωρήσουμε στο στόχο 5 των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Όσο σκιώδης, η Κλέρ θέλει να υπογραμμιστεί το μήνυμα τις εισηγητρίες, γι' αυτό και υποβάλλει παραπάνω τροπολογίες για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και για να περιοριστούν και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που σίγουρα επιδεινώνουν τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών. Τονίζεται η σημασία που έχει η δημιουργία θέσης απασχόλησης για τους περισσότερους ευάλωτους και τονίζεται και η στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των συνεταιρισμών των γυναικείων. Οπότε ευχαριστεί η κλερτινή την για την γνωμοδότηση αυτή και περιμένει να οριστικοποιηθεί. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κυρία Χανιμπολ, τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τον λόγο. Καλημέρα. Ρίκο Βάρτσας ονομάζομαι και είμαι εδώ ε, εκ μέρου τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι επικοδομητικέ τροπολογίε που έχει υποβάλει η Επιτροπή σα. Μερικά πραγματάκια από αυτά που άκουσα. Άκουσα ότι στηρίζεται περισσότερο το θέμα της συνεκτίμησης του φίλου αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της πρόταση θέσπιση του Μηχανισμού Γειτονία Ανάπτυξη και διεθνού Συνεργασία του ΝΤΙΤΣΙ. Φυσικά και θέλουμε να προωθήσουμε την ισότητα μεταξύ άλλων και στα δικαιώματα τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές μπαίνει στις χώρες μέλη και η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι με προγράμματα στις χώρες μέλη ακριβώς για να εστερνιστούν αυτό το θέμα και οι χώρες μέλη. Εμείς αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και φυσικά και προσβλέπουμε στις επόμενες συζητήσεις που θα γίνουν για αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Τώρα στην κυρία Φορέντσα θα δώσω το λόγο πάλι, στην εισηγήτρια. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις παρεμβάσεις νωρίτερα το πρωί. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους σκιώδεις. Να επιστε... προσθέσω απλόν ότι ο στόχος υπερθμών 5 για το gender mainstreaming είναι κάτι που πλαισιώνει αν θέλετε όλη μας την προσπάθεια ε, σχετικά με την σεξουαλική υγεία πιστεύω ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας ε, δεν θα πρέπει να υποβιβάζεται ή μάλλον να ε, αν να προσανατολίζεται από τα όσα λείπουν από, άλλες, από τη δουλειά άλλων επιτροπών. Νομίζω ότι το δικό μας αντικείμενο είναι να ονοματίζουμε τέτοιου είδους θέματα όπως η σεξουαλική υγεία, όπως η ελεύθερη επιλογή ω κεντρικά ζητήματα και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Και πιστεύω ότι είναι και καθήκον της Επιτροπής μας, που ασχολείται με τα θέματα ισότητα, να μην διακρίνει μεταξύ νομίμων ή όχι μεταναστών, αλλά να διαφυλάτει τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ανθρώπων νομίζω ότι και κατά την ψήφιση μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much, Ms. Ευχαριστούμε πολύ την Ελεονόρα Φορέντσα. «27 Νοεμβρίου θα γίνει ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή μας. Before I get uh, so small, a few minutes break, okay? Θα διακόψουμε για λίγα λεπτά, έτσι, στις 11 θα αρχίσουμε, αλλά καλύτερα νωρίτερα να έρθουμε. Τι θέλετε, για τα τώρα, στις 11, ωραία, 11 θα επανέλθουμε. Παιδιά θύματα ή μάρτυρες ενδοικογενειακής βίας με βάση το φύλλο. Είναι η ακρόασή μας. Αρχίζουμε με την ακρόασή μας. Είμαστε στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για παιδιά, θύματα ή μάρτυρες ενδοικογενειακής βίας με βάση το φύλλο. Πρώτα απ' όλα θέλω να καλωσορίσω εδώ τους επισκέπτες μας από την Ισπανία που είναι συγγενείς θυμάτων ε, ενδοικογενειακής βίας. Καλώς ήρθατε. Η ενδοικογενειακή βία είναι παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών, είτε είναι τα ίδια θύματα, είτε είναι απλώς μάρτυρες ενδοικογενειακής βίας. Η ενδοικογενειακή βία έχει επιπτώσεις στην ε, παρετέρω ανάπτυξη των παιδιών. Όταν εκτίθενται σε δικογενειακή βία τα παιδιά, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν το δικαίωμα σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Η ενδοικογενειακή βία εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο στα παιδιά. Μπορεί να είναι σεξουαλική, μπορεί να είναι ψυχολογική ή φυσική βία, σωματική βία. Η Επιτροπή των Γυναικών με την ακρόαση αυτή έχει καλέσει τέσσερις εμπειρογνώμονες για να συζητήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, θύματα ή μάρτυρες ενδοοικογενειακής ε, βίας που καμιά φορά φτάνει στο σημείο να βλέπουν η μητέρα τους να σκοτώνεται από τον πατέρα τους. Θα αρχίσουμε λοιπόν με την ακρόαση αυτή και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στην κυρία Μαρίσα Σολέτο Άβυλα που είναι διευθύντρια του Ιδρύματος για τις Γυναίκες της Ισπανίας, Φουνταθιών Μουχέρες. Ευχαριστώ πολύ. Και καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ στην Επιτροπή αυτή γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μας προσκάλεσε να έρθουμε και να συμμετάσχουμε στην ακρόαση αυτή. Είμαστε μια κοινωνική οργάνωση που ονομάζεται Φονταθιών Μουχέρες, Ίδρυμα για τη Γυναίκα. Και θα μοιραστούμε μαζί σας τις εμπειρίες μας από το έργο μας που είναι να αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις που η ενδοικογενειακή βία έχει στα παιδιά ενδοκογενειακή βία με βάση το φύλλο. Ξέρετε ότι η Ισπανία έχει νομοθεσία, έχει ρυθμίσει το θέμα της ενδοκογενειακής βίας με βάση το φύλλο, βία που ασκούν ε, οι σύντροφοι στις γυναίκες τους και αυτό από το 2005. Και έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε καλά γιατί υπάρχουν στατιστικά δεδομένα για αυτού του είδους το φαινόμενο στην Ισπανία και έτσι γνωρίζουμε καλά ποιες είναι οι επιπτώσεις της δικογενειακής βίας. 14 χρόνια αφού το άρχισε να ισχύει η νομοθεσία αυτή, αρχίζουμε και να αναρωτιόμαστε πώς θα βελτιώσουμε την νομοθεσία αυτή και τι επιπλέον μέτρα θα έπρεπε να υιοθετήσουμε. Εγώ έρχομαι να σας πω ποια είναι τα συμπεράσματά μας όσον αφορά ε, τα παιδιά. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία, τα δεδομένα τα οποία έχουμε και που αφορούν τα παιδιά. Το πρώτο λοιπόν που έχω να σας πω είναι ότι η αρχική νομοθεσία το 2004 κατά πάσα πιθανότητα κάτι ξέχασε. Κάτι σημαντικό. Δεν έχει συμπεριλάβει σαν απευθείας θύματα της ενδοικογενειακής βίας τα παιδιά. Κάτι το οποίο έχει συνέπειες στην προστασία τους και στη δυνατότητα να προστατευτούν καλύτερα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια από την κακομεταχείριση αυτή σε βάρος της μητέρας τους. Ένα παιδί δεν αποτελεί καθαρά μάρτυρα της ενδοικογενειακής βίας. Σε πολλές περιπτώσεις στην Ισπανία τα επίσημα στοιχεία μας λένε ότι το 70% των γυναικών που δολοφονήθηκαν από ε, Του συντρόφους τους είναι γυναίκες. Δηλαδή στο 70% των περιπτώσεων υπάρχουν παιδιά και σε πολλές περιπτώσεις είναι παρόντα τα παιδιά στη δολοφονία. Σε πολλές περιπτώσεις επίσης έχουν υποφέρει και αυτά απευθείας από τη βία. Έτσι λοιπόν Στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολη τα λέει επίσης, Πάντω από το 2005 αναγνωρίζει τα παιδιά η Ισπανία, μάλλον το 2015, σαν θύματα, απευθείας θύματα της ανδικογενειακής βίας, χάρη στην σύμβαση της Κωνσταντινούπολη Τώρα, ε, με τις μελέτες που έχουμε κάνει, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το να ζει κανείς σε δικογενειακή βία επηρεάζει το χαρακτήρα και την ψυχολογία του παιδιού. Όταν υπάρχει ένα σημαντικό συμβάν, δολοφονία για παράδειγμα, ε, αυτό είναι πολύ άσχημα για το παιδί γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί πλήρως όπως θα το έκανε αν δεν ήταν μάρτυρας ενός τέτοιου βίου γεγονότος. Γι' αυτό λοιπόν και χρειάζονται μηχανισμοί που να βγάζουν το παιδί από αυτή την κατάσταση. Έχω επίσημα στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε, στατιστικά δηλαδή, στην Ισπανία. Από τότε που αρχίσαμε να καταμετρούμε τα θύματα δολοφονιών εξαιτίας της ενδοοικογενειακής βίας, έχουμε από το 2003 χίλιες γυναίκες θύματα. Τώρα για τους ε, ανήλικους που έχουν ε, δολοφονηθεί, έχουμε μόνο από το 2013, αλλά από το 2013 στην Ισπανία δολοφονήθηκαν 27 παιδιά σε καταστάτη τέτοιες ενδοικογενειακής βία σε βάρος των γυναικών. Από το 2013, 200 περίπου παιδιά έμεναν ορφανά, γιατί δολοφονήθηκε ακριβώς η μητέρα τους εξαιτία της ενδοικογενειακής βίας. Όταν ε, όμως αναλύουμε ε, στα δικαστήρια τι απάντηση δίνεται σε τέτοια γεγονότα, τι κάνει η δικαιοσύνη δηλαδή για τις οικογένειες αυτές, βλέπουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις παραμένουν ως δικαιώματα το δικαίωμα επίσκεψης ή συκιδεμονίας ε, του αλγονιού του πατέρα δηλαδή, ακόμα και αν είναι δολοφόνος, ακόμα και αν έχει καταδεκαστεί ε, χωρίς δικαίωμα έφεσης για σοβαρά εγκλήματα. Έτσι έχουμε καταστάσεις πολύ δύσκολες για τα παιδιά. Υπάρχουν οικογένειες που έπρεπε τα παιδιά των γυναικών αυτών των δολοφονημένων να είναι υποχρεωμένες να τα πηγαίνουν στη φυλακή για να επισκεφθούν τον πατέρα τους. Δεν έχουμε επίσημα στατιστικά στοιχεία, πάντως από το 2015 φαίνεται μετά από μια κοινοβουλευτική ερώτηση μιας προβουλευτού ε, Ισπανίδας των σοσιαλιστών μας είπαν ότι τουλάχιστον 40 ανήλικοι μέσα σε ένα χρόνο πήγανε στις φυλακές για να επισκεφθούν τους πατέρες τους, δολοφόνους, είτε καταδικασμένους, είτε σε προφυλάκηση. Και τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις είχαν να κάνουν με όντως δολοφονίες. Υπάρχουν ε, επίσης οι ανάδοχες οικογένειες που υποχρεούνται να πηγαίνουν τα παιδιά να συναντήσουν τον ε, πατέρα τους που κακοποίησε, δολοφόνησε τη μητέρα τους. Όλα αυτά έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη του παιδιού, στην ε, παρετέρω εξέλιξή του, γιατί οι επιπτώσεις είναι άμεσες στο παιδί. Σήμερα υπάρχουν διάφορα μέτρα που οι οργανώσεις γυναικών, το φεμινιστικό κίνημα, αλλά και οι οργανώσεις προστασίας της παιδικής ηλικίας προσπαθούν να βελτιώσουν την νομοθεσία στην Ισπανία. Ένα από τα ζητήματα που πιστεύουμε ότι είναι θεμελιώδες είναι να ξέρουμε ότι η άσκηση ενδοικογενειακής βίας είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να περιορίζει το δικαίωμα στην κυδαιμονία. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί για ανδεκογενειακή βία πρέπει να το αφαιρείται η κυδαιμονία και δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις για τη ζωή των παιδιών. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στις υπηρεσίες για την παιδική ηλικία στην Ισπανία και αυτό είναι ότι πολλές φορές όσοι έχουν καταδικαστεί δεν συμφωνούν τα παιδιά τους να έχουν ψυχολογική υποστήριξη από τις υπηρεσίες του κράτους. Γιατί ακριβώς εφόσον διατηρούν την κυδαιμονία μπορούν να απαγορεύσουν τα παιδιά τους να έχουν τέτοια ψυχολογική βοήθεια. Σήμερα λοιπόν προσπαθούμε να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις στην Ισπανία για να αποφεύγονται τέτοιες περιπτώσεις. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα τεράστιο εμπόδιο και γι' αυτό θα σας ζητήσω κάποια πράγματα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρώπη γενικότερα. Γιατί πολλά από αυτά τα ζητήματα έχουν να κάνουν με την ερμηνεία του οικογενειακού δικαίου που γίνεται πέρα από το διεθνές δίκαιο. Ευτυχώς, σε θέματα οικογενειακής βίας, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ε, δημιούργησε κάποια ομοιομορφία στην νομοθεσία στην Ευρώπη και για τα παιδιά λέει ότι το κράτος είναι υπεύθυνο να αποφύγει τον κίνδυνο από την επαφή με τους δολοφόνους. Όμως υπάρχουν και άλλες συμβάσεις διεθνείς, της Χάγης, ε, για τις επαφές με τους ανήλικους κτλ. που ισχύουν. Και ακόμα και αν δεν έχουν κυρωθεί, αποτελούν στοιχεία που επιδέχονται ερμηνεία από τα δικαστήρια και ακριβώς βάζουν ε, το, την πατρική σχέση πάνω από οτιδήποτε άλλο. Η ισπανική δικαιοσύνη, φαντάζομαι και σε άλλες χώρες, καθορίζει ότι η σχέση αυτή πατέρα-παιδιού είναι κάτι θετικό, ακόμα και αν έχει προβεί σε σοβαρό παράπτωμα ή σε έγκλημα ο πατέρας σε βάρος της μητέρας. Ξέρω ότι στα θέματα τα ποινικά δεν έχετε άμεσα αρμοδιότητα, αλλά το έχουμε κάνει και άλλη φορά και θέλουμε να ζητήσουμε να κάνετε συστάσεις στις χώρες μέλη, όχι μόνο για να υπάρχει μια ομοιομορφία στην ομοθεσία όταν πρόκειται για την ενδοικογενειακή βία, ομοιομορφία δηλαδή να υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά να γίνουν και συστάσεις από εσά σε θέματα οικογενειακού δικαίου και να αρχίσουμε να λέμε ότι όταν υπάρχει εγκληματική συμπεριφορά να λαμβάνεται υπόψη στα δικαιώματα του εγκληματία, να περιορίζονται αυτά απέναντι στα παιδιά του. Θα πρέπει επίσης οι διάφορες συμβάσεις να αναθεωρηθούν που προβλέπουν ε, με αυτή τη σχέση ε, πατέρα-παιδιού και να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα των οικογενειών αυτών που είναι αντιμέτωπες με την τραγωδία αυτή της αδικογενειακής βίας και που όμως πρέπει να προχωρήσουν προστατεύοντας τα δικαιώματα των παιδιών. Η πρόεδρος πριν ε, είπε ότι έχουμε μία ομάδα εδώ ε, οικογενειών που είχαν θύματα και θανατηφόρα μάλιστα, δολοφονίες δηλαδή, εξαιτίας δικογενειακή βία χάσανε ε, παιδιά, νύψια, ξαδέρφια. Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε και ζητούμε να γίνει μια μελέτη γιατί σε, ευρωπα... σε ευρωπαϊκό επίπεδο μελέτη. Γιατί πιστεύω ότι όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε για τι συνέπειε από την δικογενειακή βία σε βάρος των γυναικών, αυτό βέβαια είναι καλό, αλλά δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για το τι γίνεται με τα παιδιά τους, τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά σε αυτά τα παιδιά. Τι δυσκολίες επίσης αντιμετωπίζουν ε, εκείνοι οι οποίοι αναλαμβάνουν να μεγαλώσουν στη συνέχεια αυτά τα παιδιά μετά από κάποιο έγκλημα. Θα έπρεπε να υπάρχει κάποια βοήθεια για τις οικογένειες. Εμείς διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ένα σωρό διοικητικά προβλήματα κοινωνικής προστασίας κλπ. Όπως επίσης και με το θέμα αυτό της κυδαιμονίας που παραμένει στον πατέρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα προσπαθούμε σιγά σιγά να εξηγήσουμε το πρόβλημα και στις οργανώσεις που προστατεύουν τα παιδιά. Υπάρχει μια νομοθεσία που ετοιμάζεται αυτή τη χρονιά και ζητάμε η δικογενειακή βία να αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα όταν αποφασίζουμε για την προστασία των παιδιών. Και οι άντρες αυτοί οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για ενδοικογενειακή βία να μην μπορούν πια να έχουν την κυδαιμονία του παιδιού τους. Νομίζω ότι αυτό είναι ο σωστό δρόμο. Οι οικογένειε που είναι σήμερα εδώ μαζί μα μας έχουν εξηγήσει τι δυσκολίε αντιμετωπίζουν, τι προβλήματα έχουν να ξεπεράσουν όταν μεγαλώνουν αυτοί τα παιδιά ενό αδερφού, μια αδερφή. Είναι πολλά και δεν τα γνωρίζουμε πάντα. Οπότε επαναλαμβάνω αυτό που είχαμε ζητήσει και την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσει την καλύτερη γνώση του προβλήματος, να ενημερωθούν όσοι ενδιαφέρονται για αυτή την κατάσταση, για το τι συμβαίνει στις διάφορες χώρες και να προωθήσουμε και μια γενική μελέτη. Αυτά θέλουμε να είχαμε να σας πούμε. Και από εκεί πέρα είμαστε στη διάθεσή σας. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, ευχαρίστω. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην ε, δόκτωρα Σέρι από το Ίδρυμα για τις ε, μελέτες για την οικογένεια από τη Μάλτα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα στο, στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εμπειρίες αυτές ε, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και το γεγονό ότι του δίδεται σημασία πλέον. Γιατί συχνά έχουμε θύματα ενδοοικογενειακής βία, τα οποία αγνοούνται ή μένουν στο περιθώριο. Είναι σημαντικό να παρακολουθούμε αυτά τα επεισόδια. Εδώ εκπροσωπώ την φωνή των γυναικών που έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες σε ένα πλαίσιο κρουσμάτων βίας. Αυτό είναι το πεδίο, αν θέλετε, της ειδικότητάς μου. Και πέραν της ακαδημαϊκής μου ιδιότητας, Είμαι ψυχολόγος, ε, έχω ασχοληθεί με αγωγές ε, και θεραπείες ε, σε θέματα ακριβώς αντιμετώπισης κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας και αυτό είναι το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι. Έχω ξεκινήσει Έχω μάλλον προετοιμάσει μια παρουσίαση. Θα ξεκινήσω με μια παράθεση της Ανίτας, 35 ετών, που λέει σε ένα παιδί ε, Λέει μάλλον πώς θα μπορούσα να έχω μιλήσει, δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς, υπάρχει φόβος, υπάρχει τρόμος, ακόμα και μια ενήλικη γυναίκα είναι τρομοκρατημένη, πόσο μάλλον ένα παιδί που αισθάνεται ότι είναι μόνο του και ότι δεν ζει πραγματικά. Θα ήθελα επίσης να σας μιλήσω για την 43χρονη ε, Τζέσικα, η οποία υπήρξε θύμα και μάρτυρας ενδοοικογενειακής βίας. Ο πατέρας της δολοφόνησε τη μητέρα της και λέει ότι ασχολείται ε, με ένα εστιατόριο, ε, γυρνούσε στο σπίτι μεθυσμένος, αργά και απλώς για να έχει ε, σεξ, ε, σεξουαλική επαφή με την μητέρα μου. Αλλά στις 3 η ώρα τη νύχτα δεν είναι όμορφο να ξυπνάει κανείς με, τέτοιες, με τέτοια φασαρία, με τέτοια φαινόμενα, άρχισε να την κακοποιεί, να την ε, χτυπάει πολύ συχνά και στο κεφάλι χρησιμοποιώντας ε, κουτιά και άλλα αντικείμενα. Με ξυπνούσε λοιπόν μες στη νύχτα για να πάω μαζί της στην τουαλέτα γιατί ήταν τρομοκρατημένη. Δηλαδή βλέπει κανείς ότι ε, τα παιδιά αυτά δεν υπήρξαν απλώς μάρτυρες και θύματα μεμονωμένα, αλλά έχουν και τις δύο αυτές ιδιότητες. Γιατί ζουν καθημερινά με την οικογένειά τους και συμμετέχουν σε αυτά τα επεισόδια. Και πρέπει, όπως πολλοί ειδικοί λένε, να καταλαβαίνει κανείς το πλαίσιο. Υπάρχουν αλληλουχίες πιο ήμερων ή πιο καλών ημερών με πιο κακά επεισόδια βίας ή πιο επιβλαβή. Και πολύ συχνά κανείς παίρνει την πλευρά του ενός ή του άλλου. Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο. Τώρα ποια είναι η έκταση του προβλήματος. Γνωρίζουμε ότι στι ΗΠΑ περί τα 15 εκατομμύρια παιδιά είναι εκτεθειμένα και, και 7 εκατομμύρια εξ αυτών σε σοβαρά, εκτεθειμένα σε σοβαρά κρούσματα βίας. Ε, γνωρίζουμε επίσης ότι το 23% των γυναικών έχουν υπάρξει, έχουν ε, την εμπειρία σεξουαλικής ή άλλης βίας και το 73% των, παιδιών των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρουν τέτοια επεισόδια, αλλά δεν έχουμε τον, το, το μέγεθος των παιδιών συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Eurostat επεξεργάζεται μελέτες και στοιχεία από τα οποία ίσως να απορρέουν πιο συγκεκριμένα μεγέθη για τα παιδιά που είναι δηλαδή μάρτυρες ενδοοικογενειακή βίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω να έχουμε το μέγεθος. Όπως σχολίασε και η προηγούμενη ομιλήτρια. Ως προς την περιπλοκότητα του φαινομένου γνωρίζουμε από μελέτε ότι υφίσταται ε, ενδοοικογενειακή βία κατά των παιδιών με άλλου είδους καταχρήση κατά των παιδιών η επικάλυψη είναι μεταξύ του 20 και του 70% δηλαδή των παιδιών που υφίστανται βία και υφίστανται άλλου είδους καταχρήσεις. Και η Ανίτα λέει ότι ε, τη ρωτήσαμε αν αυτά ίσχυαν και όταν ήταν μικρή και μας λέει ναι, ήμουν απόλυτα τρομοκρατημένη. Το οποίο ήταν κατανοητό γιατί ο πατέρας της έδερνε, κακοποιούσε τα παιδιά διαρκώς και αυτό αφήνει σημάδια για το υπόλοιπο της ζωής, το οποίο συνέβη και με την Ανίτα, η οποία λέει ότι θυμάμαι ακόμα αυτά τα ξυλοκοπήματα, ακόμα σήμερα και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. γιατί μας αναφέρει ότι αυτή έβγαινε να αγοράσει κάποιο γλυκό και επέστρεφε στο σπίτι και την ξυλοκοπούσε ο πατέρας της γιατί δεν είχε ε, πάρει αρκετά χρήματα μαζί τη ή οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με αυτό που της είχε αναθέσει. Πάντως, παρατηρούμε τα προβλήματα και ακαδημαϊκά και τα υπόλοιπα ψυχολογικά προβλήματα που συνδέονται με τα επεισόδια αυτά, με, τα, με την συμπτωματολογία των μετατραυματικών δηλαδή διαταραχών, το PTSD, Επίσης έχουμε υπερενεργητικότητα, ε, έχουμε bullying, δηλαδή έχουμε μια άσκηση έμεσης βίας, ψυχολογικής βίας, που συνδέονται με τα επεισόδια αυτά. Γιατί πολύ συχνά έχουμε ε, καταγγελίες για παιδιά που ασκούν τέτοια βία στο σχολείο, bullying ας πούμε στο σχολείο, ενώ στην πραγματικότητα είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και γι' αυτό συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο τον παραορμητικό που συμπεριφέρονται. Οι μελέτες μας δείχνουν ότι παρότι πολλά από τα παιδιά έχουν υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας, από μελέτη του 2006 ε, διαβάζουμε σχετικά με ένα ε, φαινόμενο που ονομάζεται sleeper effect, είναι το φαινόμενο δηλαδή της πυθούς που ασκείται προς τα παιδιά και που αυξάνει το επίπεδο Τη βία σύν το χρόνο, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ανθεκτικότητά τους. Εδώ έχω και εγώ κάνει συγκεκριμένη έρευνα σχετικά με τον τριγωνισμό, όταν δηλαδή κανείς συμμετέχει στους τσακωμούς μεταξύ των γονιών του και λαμβάνει την θέση του ενός ή του άλλου. Αυτά τα φαινόμενα δεν σταματούν όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, ενηλικιώνονται και φεύγουν από το σπίτι. Αντιμετωπίζεται δυσκολία με τα με τις ε, συναισθηματικές αντιδράσεις, τον θυμό, την οργή. Υπάρχουν δηλαδή επιπτώσεις που πρέπει κανείς να τις μελετήσει και κάτι που μας ρωτούν διαρκώς είναι κατά πόσον τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας έχουν αυξημένο κίνδυνο να γίνουν θύτες στο μέλλον. Παρότι είναι ένας υψηλός παράγοντας κινδύνου η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι παράγοντας, αναγκαστικός και υποχρεωτικός παράγοντας άσκησης βίας από το, τους ανθρώπους αυτούς στο μέλλον. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να οδηγηθούν στην άσκηση της βίας οι ίδιοι, τα ίδια τα θύματα. Δεν είναι μια κατάσταση που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ή να αλλάξουν. Η πρώιμη εγκατάλειψη των σχολείων από τα παιδιά ή η χρήση ναρκωτικών ουσιών συνδέονται με την άσκηση βίας αντιθέτως και νομίζω ότι αυτές είναι οι περιοχές στις οποίες πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Χρειάζεται λοιπόν μια ισχυρή σχέση ε, στην οικογένεια. Ε, εδώ είναι οι δείκτες και οι παράγοντες που πρέπει να επεξεργαστούμε χρειάζεται υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της εφηβείας, ένα θετικό κλίμα στο σχολείο, μια καλή σχέση με τους δασκάλους, μια καλή αποδοχή από τους φίλους, την παρέα, την κοινωνία δηλαδή των μαθητών. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω να επενδύσουμε ως Ευρωαϊκή Ένωση λοιπόν σε συγκεκριμένες μελέτες που θα μας δώσουν τα ακριβή μεγέθη σε όλα αυτά. Πρέπει να ε, εργαστούμε στην αποτροπή της ενδοοικογενειακής βίας σε όλο τον κύκλο της ζωής. Συνεργαζόμαστε με τον ΠΟΗ και τα Ηνωμένα Έθνη. Γνωρίζουμε στρατηγικές που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και που έχει αποδειχθεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές στην πρόληψη της ε, ενδοοικογενειακής βίας. Χρειάζεται έγκαιρη διάγνωση, χρειάζεται screening Εντοπισμό ε, τέτοιων επεισοδίων και φαινομένων έγκαιρα. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε τους άνδρες και να εργαζόμαστε και μαζί τους, να συνεργαζόμαστε μαζί τους ως πατέρες, αλλά και ως ανθρώπους που μπορεί να έχουν ε, κακοποιήσει τις συντρόφους τους. για η διακριτή αλλά και από κοινού μελέτη θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην πιο επιτυχή αποκατάσταση κοινωνικά και οικογενειακά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Σάντι Πλάτζετ, η οποία είναι διευθύντρια της UNICEF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 θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω ε, ζητώντας σας να θυμηθείτε μία εποχή, τότε που ήσασταν εσείς παιδιά. Ποιο ήταν το κέντρο της ε, ζωής σας, αν υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα, σε ποιον στροφόσασταν, όταν ε, πληγωνόσασταν, σε ποιον πηγαίνατε, στην οικογένεια και στο σπίτι σας. Κάθε παιδί χρειάζεται ένα ασφαλές σπίτι χωρίς βία με γονείς που το αγαπούν και το προστατεύουν. Όταν ε, τα πράγματα πηγαίνουν στραβά έξω, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο σπίτι, σε ένα, ε, σε ένα χώρο υποστήριξης. Αυτό ε, αναφέρεται στην Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού που έχει επικαιρωθεί από όλες τις χώρες του πλανήτη πέραν μίας. Όμως γνωρίζουμε και ακούσαμε μαρτυρίες ότι υπερβολικά πολλά παιδιά ε, το σπίτι τους δεν είναι ένας ασφαλής παράδεισος. Οπότε ε, τα δεδομένα είναι δύσκολα διότι τα, ε, τα η ενδοικογενειακή βία αποτελεί κατάφορη παραβίαση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γνωρίζουμε ότι εκατοντάδε εκατομμύρια παιδιά εκτίθενται στην ενδοκινιακή βία. Υπολογίζουμε ότι περίπου στα 300 εκατομμύρια παιδιά ηλικία 2 έω 4, δηλαδή πολύ νέα παιδιά, βιώνουν ε, βίαιη ε, συμπεριφορά από τους γονείς τους και παρόλα αυτά παγκοσμίω 176 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ζουν με τις μητέρες τους που είναι ε, θύματα βίας από τον σύντροφό τους και όπως σας είπα η ενδοκιγενειακή βία και η φιλετική βία κατά των γυναικών συνδέεται άμεσα ε, με την ε, βία κατά των παιδιών και φυσικά αυτό έχει ε, σοβαρή επιρροή στη ζωή των παιδιών και παρά τις σημαντικές συνέπειες στα παιδιά και τις οικογένειες αυτό φέρει ένα σημαντικό κόστος στις χώρες και στις κοινωνίες. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η ενδοκυγενειακή βία κατά των γυναικών και των παιδιών δεν περιορίζεται μονάχα σε κάποιες χώρες ή υπήρους, δεν περιορίζεται σε εθνικότητες, θρησκείες, ε, κοινωνικό-οικονομικό στάτους. Είναι ένα παγκόσμιο ε, φαινόμενο το οποίο ε, διέπει όλες τις κοινωνίες. Τώρα όσον αφορά τη βία κατά των παιδιών θα ήθελα να επαναλάβω κάποια από τα πράγματα τα οποία προαναφέρθηκαν και ισχύει ότι και ισχύουν είτε επηρεάζουν τα παιδιά άμεσα ή έμεσα. Στα βρέφη και τα μικρά παιδιά τα οποία εκτίθενται σε ενδοοικογενειακή βία βιώνουν τόσο εντονό συναισθηματικό στρες το οποίο μπορεί να επηρεάσει την σωματική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη ο εγκέφαλός τους επηρεάζεται ε, και η γνωστική τους ανάπτυξη ε, βλάπτεται αυτό έχει δραματικές συνέπειες λοιπόν και το υπόλοιπο της ζωής τους. Δεν είναι κάτι λοιπόν το οποίο περιορίζεται χρονικά. Γνωρίζουμε ότι η βία επηρεάζει τις μαθησιακές ε, ικανότητες και αποδόσεις στο σχολείο. Μία έρευνα έδειξε ότι το 40% των παιδιών που εκτίθενται στη βία έχουν χαμηλότερες αναγνωστικές ικανότητες από ότι ε, παιδιά από μη βία περιβάλλοντα. Το οποίο σημαίνει ότι στο μέλλον τα παιδιά αυτά και οι έφηβοι αυτοί θα έχουν λιγότερες εργασιακές δυνατότητες, οικονομική αυτονομία, και κατ' επέκταση θα κινδυνεύουν περισσότερο να υποπέσουν σε καθεστώ ένδυα. Επίση, αυξάνονται οι πιθανότητε κατάθλιψη ασθενειών ακοινωνικών συμπεριφορών ε, και κινδυνεύουν έτσι περισσότερο ε, να κάνουν χρήση ναρκωτικών, να επιδείξουν παράνομες παραβατικές συμπεριφορές, ε, έχουν προβλήματα να κάνουν φίλους, να κοινωνικοποιηθούν και τα παιδιά αυτά που εκτίθενται σε βία έχουν πιο επιθετική συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα σχολικό εκφοβισμό και είναι τρεις φορές πιο πιθανό να μπλέξουν σε Τα αγόρια και τα κορίτσια αντιδρούν με διαφορετικούς τρόπους. Τα κορίτσια εσωτερικοποιούν την βία αυτή σε μία από τις έρευνές μας έχουμε δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι περίπου το 50% των κοριτσιών 15 με 19 χρονών παγκοσμίω θεωρούν ότι ο σύζυγος μερικές φορές ε, δικαιολογείται που, που χτυπά την γυναίκα του για τα αγόρια από την άλλη μεγαλώνουν ε, με ένα μοντέλο τοξικής αρνοπότητας το οποίο τους οδηγεί να αναπαράγουν αυτήν την ε, βία προς τις γυναίκες. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Ε, θα πρέπει να τονίσουμε το κατεπήγον όμως του θέματος. Ε, θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται ε, για μια παγκόσμια, ευρωπαϊκή, εθνική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Θα πρέπει να αποφύγουμε κάθε τέτοιο φαινόμενο, διότι εφόσον έχει συμβεί, τα παιδιά αντέχουν και μπορούν να ξεπεράσουν παρόλα αυτά όμως έχουν περάσει ένα βαθύ τραύμα. Οπότε η πρόληψη είναι το σημαντικό. Ε, εκστρατείες, ε, σεμινάρια ε, για τους γονείς θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, προσβάσιμα για όλους, άνδρες, γυναίκες αγόρια κορίτσια, ούτως ώστε να καταλάβουν ότι είναι κάτι λάθο η χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας απέναντι στα παιδιά είναι κάτι λάθο και ότι υπάρχουν εναλλακτικέ στη χρήση βίας, διότι πολλές φορές ε, συναντάμε γονείς που οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι άλλο μπορούν να κάνουν πέρα του να ουρλιάξουν ή να χτυπήσουν τα παιδιά τους. Επίσης θα πρέπει να ξέρουν οι ενήλικες ότι υπάρχουν νομικές κυρώσεις για τους ε, θήτες, οπότε ε, από αυτό το σημείο το παιδί παίζει σημαντικό ρόλο για να σταματήσουμε τον κύκλο της βίας. Από μικρή ηλικία τα παιδιά θα πρέπει να έχουν εναλλακτικά πρότυπα όταν υπάρχει βία στο σπίτι και εδώ τα σχολεία έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο έχουμε υποστηρικτικά προγράμματα στα σχολεία που μπορούν να ε, αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο, βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν θετικές ε, στάσεις και συμπεριφορές και να αναπτύξουν ε, δεξιότητες ώστε να αποφεύγουν τέτοιες συμπεριφορές. Επίσης θα πρέπει να ενημερώσουμε για το θέμα της ενδοικογενειακής βίας, όπως για παράδειγμα την επιρροή που έχει στα παιδιά. Και φυσικά θα πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτό το θέμα. Η ενδοκιογενειακή βία δεν είναι κάτι το οποίο λαμβάνει χώρα μέσα σε τέσσερις τείχους και είναι ένα πρόβλημα μονάχα της οικογένειας. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Ολόκληρη η κοινωνία θα πρέπει να ενημερωθεί για αυτό. Οπότε οι ε, προστατευτικέ πολιτικές τη κυβέρνηση θα πρέπει να συνάδουν ε, με προσπάθειες αλλαγής συμπεριφορές και όσο δεν μιλάμε για αυτό το θέμα τόσο θα συνεχίζεται. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε επίση στις ε, φιλετικές νόρμες διότι αυτές βοηθούν στο να συνεχίζεται η βία. Γνωρίζουμε ότι επηρεάζει κυρίω γυναίκε και κορίτσια και γι' αυτό το λόγο οι διοκτικέ αρχέ. Ε, η κοινωνική λειτουργή, το προσωπικό υγεία ε, θα πρέπει να έχουν την αντίστοιχη κατάρτιση. Και αγόρια και κορίτσια, άνδρε, γυναίκε θα πρέπει να μάθουν ότι οποιαδήποτε μορφή βία προ οποιοδήποτε άνθρωπο είναι κάτι απαράδεκτο ασχέτω του φίλου ή τη ηλικία τα παιδιά θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι μόνα τους και έχουμε ακούσει ε, τις μαρτύριες, θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχουν ελληλίκες οι οποίοι νοιάζονται και θα τα προστατεύσουν και αυτό σημαίνει δάσκαλοι, κοινωνική λειτουργή, ε, ιατρικό προσωπικό, συγγενείς και μερικές φορές και ίσως ένας από τους γονείς αυτοί οι ενήλικες θα πρέπει να έχουν τις δεξιότητες να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τις ε, ανάγκες των παιδιών που έχουν εκτεθεί σε τέτοιες βίες και να ε, πηγαίνουν στις αντίστοιχε υπηρεσίες. Οπότε περνάμε στην ύπαρξη των υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι οριστικές και πραγματικά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του παιδιού. Το παιδί λοιπόν δεν μπορεί να πάει από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Δεν μπορούμε να ε, ε, περιμένουμε ε, από έφηβους ή από παιδιά να έχουν την δυνατότητα να πάρουν αυτή την πρωτοβουλία ούτω ώστε να πάνε από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο επαφή το οποίο στη συνέχεια θα συνοδεύει το παιδί σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες. Και οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε παιδιού. Υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες, οπότε θα πρέπει να είναι ευέλικτα. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε τις χώρες να ενισχύσουν το νομικό πλαίσιο για την προστασία των παιδιών από τις διάφορες μορφές βίας. Είναι σοκαριστικό το ότι σήμερα μονάχα 60 χώρες έχουν υιοθετήσει νομοθεσίας που αποτρέπει, ε, απαγορεύει την χρήση σωματικής βίας στο σπίτι, το οποίο σημαίνει ότι πάνω από 600 εκατομμύρια παιδιά ε, κάτω από 5 ε, δεν έχουν καμία νομική προστασία και υπάρχουν ακόμα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αποτρέπουν την χρήση βίας από τους γονείς. Οπότε η ποινικοποίηση της ενδοκογενειακής βίας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η βία δεν είναι κάτι το απαράδεκτο δεν μιλάμε το να βάλουμε τους γονείς στις φυλακές επειδή χαστούκησαν το παιδί τους οι γονεί ε, χρειάζονται ε, δεξιότητες και υποστήριξη ούτω ώστε να αποφεύγουν τέτοιε συμπεριφερές. Ε, όμως η Σουηδία για παράδειγμα έχει δείξει ότι όταν η ενδοκογενειακή βία και η βία κατά των παιδιών ποινικοποιείται τότε υπάρχει μια αλλαγή στις κοινωνικέ νόρμες. Επίση, καλούμε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ε, για την ενδοοικογενειακή βία και τη βία κατά των γυναικών και τέλος θα πρέπει να επενδύσουμε σε δεδομένα. Όπως είπα, δεν έχουμε αρκετά δεδομένα διότι το πρόβλημα αυτό παραμένει κρυμμένο μέσα στα σπίτια. Θα πρέπει να συλλέξουμε όμω αυτά τα δεδομένα για τι γυναίκε και τα παιδιά που είναι θύματα ενδοκινιακή βία. Υπάρχουν κάποιε χώρε που δεν έχουν καθόλου δεδομένα. Οπότε η επένδυση σε δεδομένα όπω είναι η συλλογή, ε, διανομή, ανάλυση, ε, χρήση θα είναι σημαντικά για την ε, διαδικασία παρακολούθηση και επίση θα τονίζει το ζήτημα τη ευθύνη που έχουν οι εθνικέ αρχέ και η διεθνή κοινότητα. Και εδώ ελπίζουμε ότι οι ε, βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι θα βοηθήσουν ε, διότι αναφέρονται επίσης και στο ζήτημα της ενδοκινητική βίας και της βίας κατά των παιδιών σε τρεις στόχους και τονίζουν ε, τη χρήση δεδομένων. Θα πρέπει να προστατεύουμε τα παιδιά, το οποίο είναι ένα μονοπάτι προς μια πιο ειρηνική κοινωνία, κάτι το οποίο ορίζεται από τον στόχο νούμερο 16 και για αυτό θα χρειαστούν μεμονωμένες και συλλογικέ δράσει για να διορθώσουμε αυτό το παγκόσμιο λάθος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σάντι Μπλανσέτ. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Πιερή Βεροσέ, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος για τα δικαιώματα του παιδιού. Είναι εκπρόσωπο τη Γαλλόφωνη κοινότητα ε, του Βελγίου. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να έρθω να σας μιλήσω για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για το δικό μου το έργο που είμαι επιτετραμένος για τα θέματα ε, δικαιωμάτων του παιδιού. Πρόκειται για έναν εξάρτητο θεσμικό όργανο που προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών στην ε, γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, στο γαλλόφωνο Βέλγιο δηλαδή. Όταν μου είπανε να σας μιλήσω για αυτό το θέμα, σκέφτηκα, μα δεν υπάρχουν πολλά. Υπάρχει το ηθικό, το σεξουαλικό, υπάρχει ο δημόσιος χώρος, η οικογένεια, η οικογενειακή βία, γι' αυτό μιλάμε. Υπάρχουν οι καταναγκαστικοί γάμοι, ο ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, καταναγκαστική εργασία κλπ. κλπ. Οπότε εννοείται, δεν είμαι πυρογνώμων για όλα αυτά. Θα επικεντρωθώ λοιπόν μόνο στην οικογενειακή βία και πολύ χάρηκα που άκουσα και την εκπρόσωπο της UNICEF για τα θέματα της βίας σε σχέση με την εκπαίδευση. Γιατί το να λέμε, ε, να χρειάζεται ακόμα σήμερα να λέμε ότι δεν κάνει καλό στο παιδί να το χτυπάμε, ε, μου φαίνεται τρομερό. Γιατί λοιπόν υπάρχει τέτοια βία και γιατί υπάρχει και η ενδοικογενειακή βία, γιατί θεωρείται κάτι τετριμένο μερικές φορές η ενδοικογενειακή βία. Είπαμε ότι τα παιδιά που εκτίθενται σε αυτή τη βία ε, πρόκειται για παιδιά είτε θύματα είτε μάρτυρες. Η βία τι επιπτώσει έχει, το ακούσαμε πολύ καλά. Εγώ όμως θα σας μιλήσω για κάτι άλλο, για το πλαίσιο. Χρειάζεται ένα δομημένο πλαίσιο το παιδί για να μεγαλώσει, που να του προσφέρει ασφάλεια. Η ενδοικογενειακή βία λοιπόν ενέχει τραυματικά για το παιδί επεισόδια, που το τρομάζουν και δεν του προσφέρουν ασφάλεια για την καθημερινή του ρουτίνα. Το παιδί χάνει επίσης και τη θέση του παιδιού, γιατί ο γονιός που εμπλέκεται σε έναν κύκλο βίας, δικογενικής βίας, δεν θα μπορέσει να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του ως γονιός. Οπότε τελικά θα αφήσει το παιδί να είναι είτε το παιδί ασπίδα, είτε το παιδί στο οποίο θα μιλάει και θα τον χρησιμοποιεί σαν φίλο θα είναι το παιδί που θα αναλάβει το ρόλο του γονιού δηλαδή μερικές φορές. Έτσι καταστρέφουμε την παιδική καθημερινότητα και δημιουργούμε τραύματα ψυχολογικά, αλλά ακόμα όπως είπαμε και μαθησιακά. Εμείς λοιπόν για την προστασία των παιδιών δημιουργήσαμε μία διατομιακή ομάδα εργασίας για το θέμα της ενδοικογενικής βίας και τις επιπτώσεις της στα παιδιά και καταλήξαμε σε ένα συμπόσιο το 2010 Εκεί συζητήσαμε τις πρακτικές δυσκολίες και προσπαθήσαμε να κάνουμε συγκεκριμένες συστάσεις. Για αυτές θα σας μιλήσω. Όλοι γνωρίζετε ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να εντοπίσουμε ότι υπάρχει ενδοικογενειακή βία και να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε έναν συζυγικό καυγά με την ενδοικογενειακή βία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στην ενδοικογενειακή βία υπάρχει θέμα ότι κάποιος κυριαρχεί εκεί πάνω σε κάποιον άλλον. Τι συνοδευτικά μέτρα μπορούμε λοιπόν να έχουμε και προς το συμφέρον πιανού, του παιδιού, της μητέρας που είναι συνήθως το θύμα, για την οικογένεια ολόκληρη. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέσαμε τότε. Οπότε οι συστάσεις μας του 2010 εξακολουθούν δυστυχώς να είναι επίκαιρες. Θέλουμε να προωθήσουμε τη δουλειά που γίνεται μέσα σε δίκτυα. Να ξέρουμε ποια είναι η αποστολή του καθενός και ποια είναι τα όρια αυτής της αποστολής για να συντονιστούμε καλύτερα. Έπειτα πρέπει να καταρτιστούν οι επαγγελματίες. Πρώτα απ' όλα να κάνουν τη διάκριση για το τι βία υπάρχει και έπειτα να αποφασίσουν τι στρατηγική θα ακολουθήσουν απέναντι στα παιδιά θύματα. Η παρακολούθηση πρέπει να είναι συνεχής. Υπάρχει και αστυνομία που έχει και αυτή ένα ρόλο να βοηθήσει τα θύματα. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας τα πρωτόκολλα συνεργασίας που υπάρχουν, γιατί ναι μεν υπάρχουν, αλλά δεν είναι γνωστά πάντα. Και να γίνουν και συγκριτικές μελέτες. Αν ε, συλλέγουμε στοιχεία τα οποία έχουν αναλυθεί, μπορούμε καλύτερα να καταλάβουμε τι σημαίνει και να σταθμίσουμε καλύτερα τις πολιτικές. Τώρα όταν μιλάμε για δημόσιες πολιτικές, μιλάμε συνήθως για μια στρατηγική. Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ενδοικογενειακής βίας. Ωραία. Υπάρχουν προγράμματα δράση σε τοπικό επίπεδο επίση. Όμω εκεί που χρειάζεται είναι το άρθρο 12 τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού που μιλάνε για τη συμμετοχή των παιδιών. Δηλαδή τα παιδιά εποφελούνται από τι δημόσιε πολιτικέ. Πώ θα σταθμίσουμε καλύτερα τι είναι καλύτερο για το παιδί. Πρέπει να ακούμε το ίδιο το παιδί τι έχει να πει. Πολλέ φορέ το λέμε στι διασκέψεις. Γιατί το να ακούσω κάποιο κύριο μια κυρία να λένε εγώ ξέρω τι είναι καλό για το παιδί και εγώ θα σας φτιάξω το κατάλληλο πρόγραμμα ε, όχι. Πώ μπορείτε να το ξέρετε. Άμα δεν με ξέρετε, μπορείτε να κάνετε ένα πρόγραμμα για μένα. Όχι. Το ίδιο ισχύει και για το παιδί, λοιπόν. Το να λέμε στο παιδί ότι είναι για το καλό σου, δεν φτάνει. Πρέπει να ακούμε το παιδί. Ποια είναι η δικιά του γνώμη. Και αυτό κάνουμε σε αυτή την ε, στρατηγική και στην αρχή στην εκπόνηση της στρατηγικής και στον έλεγχο και στην αξιολόγηση της κάθε πολιτικής. Μιλάμε λοιπόν για δημόσιες πολιτικές, οι οποίες δημιουργούνται έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη μας τις υποχρέσεις που απορρέουν από διάφορες συμβάσει όπως είναι εκείνη της Κωνσταντινούπολης. Στο Βέλιο πιο συγκεκριμένα έχουμε το πρόγραμμα δράσης μας με κατά προτεραιότητα άξονες, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, όμως οι άξονες αυτοί μιλάνε για την εκπαίδευση, για την συνδυτοποίηση μετά για την συνέχεια, την έρευνα, πώς δηλαδή θα διασφαλίσουμε την προστασία του θύματος και υπάρχει και το θέμα της συνεκτίμησης του φύλου που και αυτό λαμβάνεται υπόψη. Είναι μια σύσταση πολύ σημαντική όταν έχουμε να κάνουμε με το άσυλο και τη μετανάστευση. Η συνεκτίμηση του φύλου λοιπόν. Υπάρχουν επίσης τα άρθρα 22, 23 και 26 που μιλούν για την υποδοχή και τις συμβουλές. Εδώ πραγματικά οι χώρε στους οποίους υποδεχόμαστε τα παιδιά θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να το υποδέχονται καταρτισμένοι ενήλικες που να διαθέτουν παιδαγωγικά μέσα και να χρησιμοποιούν και μια ρητορική που να είναι κατάλληλη για τα παιδιά. Και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε με διάφορους μηχανισμούς που δημιουργούμε. Επίσης, για τις δημόσιες πολιτικές και για τη συνέχεια που δίνεται σε εγκληματικέ πράξεις. Έχουμε φυσικά την δικαιοσύνη που έχει ήδη εξετάσει το θέμα της αδικογενειακής βίας. Αναθεωρήθηκε η στρατηγική τους για να έχουμε μια στρατηγική η οποία επικεντρώνεται περισσότερο στο παιδί. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια μήνυση, πώς την ε, καταχωρούμε εμείς πώς γίνεται, μέσα από ποια διαδικασία φτάνει σε μας. Και τι γίνεται με το παιδί, τι γίνεται με το δικαίωμα στη επίσκεψη του άλλου γονιού. Ο δικαστής, ο οποίος είναι αρμόδιος για τα οικογενειακά θέματα, θα θέσει το ερώτημα. Είναι θύμα το παιδί. Πρέπει να έχει επαφές με τον πατέρα που είναι ο δράστης, ο θήτης. Αυτό όμως πρέπει να το δούμε με το συγκεκριμένο παιδί και τη συγκεκριμένη οικογενειακή του κατάσταση. Γι' αυτό πολλές φορές χρειάζεται μια διαμεσολάβηση. Προσοχή όμως μην κάνουμε το παιδί διπλά θύμα και μην του διονίζουμε το τραύμα. Πάντα λοιπόν πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικέ και να ακούμε το παιδί τι έχει να πει για τη σχέση του με τον πατέρα φίτη. Έπειτα, η προστασία μπορεί να υπάρχει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Από το 2012 μπορεί να ζητηθεί απομάκρυνση από τον πατέρα ακριβώ για να προστατευτεί η υπόλοιπη οικογένεια. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να πούμε ότι στο Βέλγιο, κυρίως στην Βαλονία, έχουμε τα λεγόμενα καταφύγια, για γυναίκες, θύματα δικογενειακής βίας και για παιδιά. Νομίζω ότι έχουμε 19 τώρα που επιδοτούνται. Εδώ βέβαια τίθεται πάλι το ερώτημα, γιατί οι γυναίκες οι οποίες θεωρείται ότι είναι σε παράνομη εντό εισαγωγικών ε, διαμονή, δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα καταφύγια. Εγώ δεν συμφωνώ με τον όρο παράνομη, έτσι. Όμως υπάρχει εμποδίζεται η πρόσβαση ε, στα άτομα αυτά, σε αυτά τα καταφύγια, ενώ δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε οποιοδήποτε παιδί, οποιοδήποτε γυναίκα να μπορεί να πάει ε, σε μια υπηρεσία. Αλλά αυτό θα το κάνει μόνο όταν είναι ενημερωμένη και γνωρίζει ότι υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν. Το παιδί, λοιπόν, είπαμε πρέπει να είναι στην καρδιά της διαδικασίας, στον πυρήνα και της δικαστικής ε, διαδικασίας να ε, το συναντάει ο δικαστής και να το ενημερώνει το παιδί και να το ακούει κυρίως. Στο Βέλγιο υπάρχουν κάποιες εντάξεις που λένε όταν είναι κάτω των 12 ε, το παιδί δεν μπορεί να πει την άποψή του. Αυτό δεν ισχύει. Διότι ναι, μένα, από τα 12 και μετά υποχρεωτικά παίρνει ένα έντυπο το οποίο πρέπει να συμπληρώσει το παιδί, αλλά και πριν τα 12 μπορεί κάλλιστα, εφόσον το ζητήσει, να έρθει σε επαφή με τον δικαστή. Θα έρθω τώρα και σε μια άλλη πτυχή, γιατί αναφερθήκαμε στην οδικογενειακή βία με βάση το φύλλο. Εδώ υπάρχει το θέμα και της ταυτότητας του φύλου και πώς εκφράζεται αυτό το φύλο. Πρέπει να σεβόμαστε το παιδί και την ελευθερία έκφρασής του. Στο Βέλγιο, σε εμά τουλάχιστον, στη δικιά μας επιτροπή, πολλές φορές ακούμε ότι δεν γίνεται σεβαστή η ταυτότητα του φύλου. Η επιλογή αν θα πάει σε ένα καταφύγιο ένα γόρι, ένα κορίτσι, ε, από αυτό θα εξαρτηθεί και η ψυχαγωγία του. Εντάξει, δεν σας μαθαίνω τίποτα ότι τα παιδιά, τα γόρια θα πάνε στο ποδόσφαιρο. Ε, το βλέπετε αυτό και στα μαγαζιά παιχνιδιών ότι υπάρχει αυτή η διάκριση για τα γόρια και τα κορίτσια. Υπάρχει ο αθλητισμός, υπάρχουν ε, τα βεστιάρια που αλλάζουν τα παιδιά. Τελικά ε, κλείνουμε το παιδί μέσα στο φίλο του. Ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις ε, των ε, ΛΟΕΔ που δεν μπορούν να κλειστούν μέσα σε ένα τέτοιο κουτί. Και είναι σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί εμείς είμαστε ένα οργανισμός στον οποίο φτάνουν προσφυγές και μας έρχονται πολλές που μας λένε ότι στο ένα ή στο άλλο πρόγραμμα για δραστηριότητες στις διακοπές οι γονείς υποχρεώνουν το παιδί να πάει και να κάνει μία δραστηριότητα η οποία θεωρούν ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στο φίλο του. Επίσης, μιλήσαμε για την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση, φυσικά και χρειάζεται η κατάρτιση. Γιατί όταν υπάρχει, υπάρχουν κάποιες νομικές διατάξεις, εννοείται ότι θα πρέπει οι αρμόδιοι να είναι ενήμεροι και πρέπει να υπάρχει και ευαισθητοποίηση στην κοινή γνώμη αλλά και στα παιδιά που είναι πολύ μικρά. Έχουμε τέτοια μαθήματα που πολύ νωρίς μπορούμε να μάθουμε τα παιδιά. Εδώ υπάρχει η ποικιλομορφία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να μάθουμε ακριβώς τα παιδιά ότι αυτή η ποικιλομορφία είναι πλούτος και πρέπει να μάθουμε στα παιδιά τι σημαίνει η διάκριση και η μη διάκριση και να καταργήσουμε την εκπαιδευτική βία που χρησιμοποιείται καμιά φορά και δημιουργεί μία σχέση κυριαρχίας του ενός πάνω στον άλλον. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε τον κύριο Γουσέ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στα μέλη για μια ανταλλαγή απόψεων. Η κυρία Γαρθία Πέρδη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε τα μέλη του πάνελ σας για τις παρεμβάσεις τους, τις παρουσιάσεις τους. Ε, είναι σημαντική και πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση γιατί μόνο ακούγοντας τις διάφορες μελέτες που γίνονται από τις κοινωνικές οργανώσεις, από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, είναι δυνατόν και έχουμε εμείς την πολιτική ευθύνη να υποστηριχθούν τέτοιες πρωτοβουλίες σχετικά με τα ζητήματα αυτά, γνωρίζοντας δηλαδή τα ζητήματα αυτά καλύτερα να ευχαριστήσω και το Ίδρυμα για τη γυναίκα και την κυρία Σολέτο. Εγνώριζα την πρωτοβουλία, της, ε, την καθόρλα δηλαδή, ε, με τις σχετικές ενισχύσεις, ε, υπογραμμίζει και περιγράφει μια πραγματικότητα που πολύ συχνά δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα της. Γιατί συχνά αναφερόμαστε για την βία μεταξύ των φίλων τη συνέχιση δηλαδή των κροσμάτων, των δολοφονιών των γυναικών, μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες, αλλά πίσω από κάθε τέτοια κρούσμα επεισόδιο υπάρχει μια ιστορία, ένα αφήγημα, ε, μια προέλευση. Και έχουμε την ευθύνη να κατενοούμε αυτές τις περιστάσεις των γυναικών που έχουν πέσει θύμα βίας γιατί μόνο έτσι θα κατανοήσουμε την πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή, τι σημαίνει από τη μία μέρα στην, στην άλλη να χάσεις έναν άνθρωπο της οικογένειάς σου, από την οικογένειά σου, έναν, έναν δικό σου άνθρωπο και τι σημαίνει αυτό από εκεί και πέρα και διοικητικά. Τι άλλο πρέπει να κάνεις από εκεί και πέρα για να το αντιμετωπίσεις, τι πρέπει να υποστείς. Νομοθετούμε λοιπόν Προσπαθούμε να κοιτάξουμε το φαινόμενο ως νομοθέτες, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική και η υπόλοιπη διάστασή του με τις παρουσιάσεις που ακούμε σήμερα. Να μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε μια ουσιαστική ανταλλαγή για να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε και την ανάπτυξη πρωτοβουλίων από των κρατών μελών, των κυβερνήσεων των χωρών. Στη χώρα μας, την περασμένη εβδομάδα, στην Ισπανία, υπευλήθη μια πρόταση νόμου ώστε να αναγνωριστεί το δικαίωμα των ενισχύσεων των ορφανών των οικογενειών, δηλαδή που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακούς φόνους και άλλη βία. Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν την κατάσταση αυτή αναλαμβάνουν το βάρος αυτό υπό οικονομικές συνθήκες κρίσεως, δύσκολες. Μιλούμε για τα... Μάλλον χρειαζόμαστε κοινωνικά συστήματα επαρκώς ευρώστα ώστε να αντιμετωπίζουν, να αναλαμβάνουν αυτές τις οικογένειες, να προσφέρουν λύσεις στα θύματα της βίας. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς υπό την οπτική γωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούμε να οθήσουμε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες και μέτρα και πώς μπορούμε να αναλάβουμε και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Αναφέρθηκαν κάποιες από τις ομιλήτριες σε σημαντικές μελέτες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να έχουμε μια ακριβέστερη χαρτογράφηση εικόνα της κατάστασης μεταξύ των κρατών μελών. Για να δούμε ποια είναι η κατάσταση και πώς μπορούμε να ανταπαγρυθούμε, να την αντιμετωπίσουμε. Γιατί μπορεί να υπάρξει και μια υποφελής επιρροή μεταξύ κρατών μελών. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε τη διενέργεια μιας μελέτης τέτοιου είδους και αν ίσως συμφωνούν και οι άλλες πολιτικές ομάδες, ίσως η συζήτηση που είχαμε σήμερα θα μπορούσε να γίνει και στην Ολομέλεια με κάποια ίσως ε, ερώτηση και προς την ε, Επιτροπή. Ξέρω ότι κινούμαστε προς το τέλος της ε, εντολής μας. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι σημαντική η πρωτοβουλία που μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ και πάλι για την συνεισφορά σας, τις παρουσιάσεις σας, τη δουλειά σας και ελπίζω να είμαστε να φανούμε στο ύψο των περιστάσεων ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σα βοηθήσουμε κι εμεί. Ευχαριστούμε την κυρία Γαρθία Πέρθ. Η κυρία Μπιόρκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους προσκεκλημένους και προσκεκλημένες. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να σας ακούσουμε. Θα ήθελα όμως ε, να αναφερθώ σε κάποια θέματα από την Σουηδική ε, Σκοπιά. Έχουμε ε, γραμμές επικοινωνίες, έχουμε οργανισμούς ε, για τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών ε, και οι οργανισμοί αυτοί όλοι είναι ξεκάθαροι για το γεγονός ότι και τα παιδιά είναι θύματα σε μια κατάσταση όπου μια γυναίκα εκτίθεται σε πατριαρχική βία. Και γι' αυτό έχουμε όλο και περισσότερα δεδομένα. Η Ισπανίδα συνάδελφος το ξεκαθάρισε αυτό βλέπ, είδαμε πριν από 15 περίπου χρόνια αυξημένες ε, αποφάσεις δικαστηρίων ε, κατά ε, πατέρων οι οποίοι παρόλο που ήταν βίαιοι κατά των συζύγων του λάμβαναν την κυδαιμονία του παιδιού ε, και πλέον όμως έχουμε μια καλύτερη κατανόηση ότι και το παιδί είναι θύμα και δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού να αναγκάζεται να περνά ε, χρόνο με κάποιον ε, ο οποίος διονύζει τη βία θύμα της οποίας είσαι. Δεν θα πρέπει να προτιμούμε τα δικαιώματα των γονέων εις βάρος των δικαιωμάτων των παιδιών τα οποία χρειάζονται προστασία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν βελτιώσεις εκεί, διότι ακόμα και στα σουηδικά δικαστήρια βλέπουμε περιπτώσεις όπου ε, χορηγούνται δικαιώματα επισκέψεις ε, ε, σε τέτοιου γονείς. Βλέπουμε ο κηδεμόνας να έχει ακόμα το δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του παιδιού παρόλο που έχει καταδικαστεί για επιβολη σε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν ε, να λαμβάνει άλλους αποφάσεις για το παιδί. Οπότε οι οργανώσεις ε, αυτές θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να διασφαλίσουν ε, για να υπάρξει μία αλλαγή η οποία δεν θα γίνει μονάχα στα χαρτιά αλλά και στην, πραγματική, στην πραγματικότητα. Επίσης υποστηρίζω τα όσα υπόθηκαν για την σωματική βία ε, ως τιμωρία ε, η Σουηδία κάνει βήματα για να απογορεύσει κάθε μορφή βίας προς τα παιδιά και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα τομέα στον οποίο θα πρέπει να εργαστούμε περαιτέρω, ε, να εργαστούμε περαιτέρω εδώ στο Κοινοβούλιο παρόλο που είναι εκτός του εύρου τη σημερινή μας ακρόασης. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη συνεισφορά σας. Εκτός μικροφώνου πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Ιχεμένες Σπάρο. Eh. Σα ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όπω και οι συνάδελφος θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ σα για την παρουσίασή του εδώ και την συνεισφορά του. Είχα κάποιες παρατηρήσεις και ίσως κάποιες ερωτήσεις να κάνω. Ε, στην ε, εφαρμογή της ε, σχετικής οδηγίας για την προστασία των δικαιωμάτων θυμάτων βίας και στην σχετική δουλειά που έχουμε κάνει για αυτήν την οδηγία υπήρχε ένα τμήμα αφιερωμένο στα παιδιά, στους ανελίκους όπως και στην βία μεταξύ των βίλων. Εκεί αποτυπωνόντουσαν δηλαδή τα παιδιά ως θύματα βίας ενδοοικογενειακής Θα ήθελα λοιπόν να κατανοήσω την άποψή σας σχετικά με το πώς αναπτύσσεται αυτή η εναρμόνιση της νομοθεσίας που είναι αρκετά δύσκολο ζητούμενο εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε διάφορα πεδία, βιομηχανικό, γεωργικό κτλ. Αλλά είναι δύσκολο να προχωρήσει η νομοθεσία διότι τα κράτη-μέλη επικαλούνται την επικουρικότητα. Και έχουμε σημαντικές διαφορές ποινικού, αστικού, κώδικα κτλ. μεταξύ της μίας και της άλλης χώρας. Όχι ότι δεν δέχονται ότι πρόκειται για ποινικά κολάσιμη πράξη, αλλά εμπίπτουν σε διάφορε άλλες ευρύτερε νομοθετικές διατάξεις. Ήθελα λοιπόν να κατανοήσω κατά πόσον θεωρείτε εσείς ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές, η άποψή μου είναι ότι δεν είναι, και στο ποια είναι η διαφορά μεταξύ των χωρών σε αυτό. Δηλαδή έχουμε δει ότι και η Ευρωπαϊκή Διαταγή για την Προστασία των Θυμάτων δεν έχει λειτουργήσει. και εκεί αναφερόμασταν στις γυναίκες που είναι θύματα ενδοκιογενειακή βίας και που ήθελαν να ζητήσουν προστασία από άλλη χώρα. Συνοδευόμενε από το ή τα παιδιά τους. Και είχαμε πάρα πολλέ τέτοιε αιτήσει προστασία Περιμέναμε πολύ μεγάλη ζήτηση και τελικώς είχαμε 7 Μιλούσαμε για δεκάδες χιλιάδων περιπτώσεις και είχαμε 7. Άρα κάτι δεν λάβαμε υπόψη μας. Ούτε η δικαστική λειτουργοί εγνώριζαν, ούτε η ΜΚΑ όμικρον, ούτε οι αστυνομικές υπηρεσίες, ούτε καν τα θύματα ότι υφίστανται αυτά τα μέσα. Επομένως η ερώτηση μου είναι τι άλλα μέσα έχουμε στη διαθέσή μας και επίσης πώς μπορεί αυτό να γίνεται γνωστό την στιγμή της καταγγελίας. Γιατί υπάρχει πολύ έντονο συναισθηματικό δεσμό, όπω είναι απολύτω φυσιολογικό μεταξύ των παιδιών και των γονέων του, ακόμα και αν οι γονεί του είναι κακοί άνθρωποι, για να το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, <clears throat> πώ μπορεί στα πλαίσια μια δικαστική εξέταση ένα παιδί να, είναι, να καταθέσει κατά του γονέα του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Χιμένεθ. Κυρία Κιάνγκε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες ε, για τις παρουσιάσεις τους και την ποιότητα των τοποθετήσεων τους. Είναι πολύ σημαντικό το σημερινό ζήτημα, ιδιαίτερα ε, σχετικά με την προστασία των ανηλίκων. Να απευθύνω ένα χαιρετισμό και στους επισκέπτες μας που προέρχονται από την Ιταλία και από ενώσεις που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προφανώς θα είναι πολύ ενημερωτική η σημερινή συζήτηση για αυτούς ε, και θα διαβιβάσουν τα μηνύματα. Έχουμε την 70η επέτειο της Χάρτας των ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και έχω την εντύπωση ότι όσο περισσότερο χρόνος ε, περνάει, τόσο περισσότερο υποχωρούν διάφορα δικαιώματα σε διάφορα μέτωπα, σε διάφορους τομείς. Επομένως, χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική επικοινωνίας, μια νέα στρατηγική ώστε να μπορέσουν οι πολίτες ε, να ξαναοραματιστούν, να ονειρευτούν. και το θέμα επίσης ε, της ε, φορητότητος, αν θέλετε να το πούμε έτσι, των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν είναι ότι κάποιος μετακινείται και πηγαίνει σε άλλη χώρα και έτσι έχει αφήσει τα δικαιώματά του εκεί που έμενε. Και βεβαίως και η εκπαίδευση και η κατάρταση που πρέπει να διέπει όλους τους φορείς με ενίσχυση των διατάξεων, αλλά χωρίς ιδιαίτερη εστίαση επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεν μπορεί κανένα τομέα και κανένα φορέα να καταλάβει περί τίνο πρόκειται και να εργαστεί αποτελεσματικά. Επομένω, μα χρειάζεται κατάρτιση από το σχολείο μέχρι του ειδικού, του εμπειρογνώμονε. Και ήθελα να μείνω για μια στιγμή, ε, καθότι εχθέ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ενεκρίθη ε, κανονισμός πολύ σημαντικός σχετικά με τα ενωσιακά στατιστικά δεδομένα. Μιλήσατε για συλλογή στατιστικών δεδομένων. Ο κανονισμός αυτός αφορά στη λογή ενωσιακών στατιστικών σε θέματα μετανάστευσης και διεθνούς προστασίας. Πρόκειται για ένα νομοθετικό φάκελο πάρα πολύ σημαντικό και το λέγω γιατί αποστέλουν πάρα πολλά στοιχεία αλλά και εις ό,τι αφορά εις τους ανηλίκους γιατί πολύ συχνά πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε επαρκή στατιστικά για τους ανήλικους. Τα κράτη-μέλη στα πλαίσια του κανονισμού αυτού θα πρέπει να βελτιώσουν την ακρίβεια και τον όγκο των δεδομένων που υποβάλλουν. Θα υπάρχει μια σειρά από υποχρεώσεις σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία και για τους ανηλίκους, επαναλαμβάνω, και γι' αυτό θέλαμε να το συμπεριλάβουμε, ιδιαίτερα για τους ε, ανηλίκους που δεν συνοδεύονται, τους ασυνόδευτους. Και σχετικά με τα νομοθετικά πλαίσια στα οποία δικαιούνται προστασίας. Γιατί εδώ έχουμε πάρα πολλά κενά και πάρα πολλές ελλείψεις και πολύ συχνά και ξεχνούμε και την φωνή, την επιθυμία δηλαδή των ανηλίκων των παιδιών, γιατί μαζί με τα παιδιά θα πρέπει και εισακούγοντας τη φωνή τους θα πρέπει να διαμορφώσουμε τα όποια νομοθετικά πλαίσια και μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση για να προχωρήσουμε και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Ζητώ συγγνώμη που με κρηγόρησα, αλλά ήθελα ε, να σας δώσω και μια μαρτυρία. Πριν από λίγα χρόνια ήμουν υπουργό ε, κοινωνικη ενταξη στην Ιταλία ε, και είχα την επίσκεψη μιας γυναίκας που ερχόταν από κάποια τρίτη χώρα γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα για τις οικογένειες της μικτές ή ξένων υπηκόων. Αυτή η κυρία λοιπόν ήταν ε, γιαγιά ενός παιδιού που, είχε, που ήταν μάρτυρας της δολοφονίας της μητέρας του και αυτή ξένη υπήκος. Ο πατέρας του Ιταλός υπήκος. Άφησαν λοιπόν το παιδί στην γιαγιά από την πλευρά του πατέρα χωρίς να σκεφτούν ότι θα μπορούσαν να το αφήσουν και στην γιαγιά της κυρίας, της ξένης. Το δικαστήριο αυτομάτως, αν θέλετε, ανέθεσε το παιδί στην προστασία της γιαγιάς της πατρικής με επίσκεψη στη φυλακή του πατέρα δηλαδή που είχε σκοτώσει τη μητέρα του μαζί με το παιδί που τα έβλεπε όλα αυτά. Εμένα μου φάνηκαν όλα αυτά τελείως παρανοϊκά και βρήκαμε μια πλατφόρμα, ένα δίκτυο δικηγόρων εκπροσώπων της ε, κοινωνίας των πολιτών. Το παιδί δεν μιλούσε. Σήμερα, μετά από δύο χρόνια, καταφέραμε να αποσπάσουμε το παιδί από την οικογένεια του πατέρα και το οποίο ζει ευτυχές με την οικογένεια της μητέρας του των λοιπόν συγγενών δηλαδή. Και άρχισε να μιλάει, άρχισε να επικοινωνεί, πηγαίνει στο σχολείο διότι η γιαγιά του παιδιού ήταν προστατευμένη και χρειάστηκε να παρέμβουμε διότι πολύ συχνά με τις μικτές οικογένειες, τα μεικτά ζευγαριά δεν λαμβάνουν υπόψη οι συνθήκες του ξένου υπηκόου που είναι το μέλος της οικογένειας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Άλισον. Αγιάλα Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ καλωσορίζω και ευχαριστώ πολύ όλους τους εισηγητές και φιλοξενούμενους μας εδώ. Αυτά που μας παρουσίασαν όντως καταδεικνύουν τις αδυναμίες και γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που επήγει και που έχει να κάνει βέβαια και με την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία. Θέλω να στηρίξω αυτά που είπατε για το ότι επήγει να υπάρξει μια συνολική μελέτη όπου να φαίνεται ξεκάθαρα ποια είναι τα θύματα της ενδοικογενειακής ε, βίας και να συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά εκτός από τις γυναίκες. και να δούμε πέρα από τα σκάνδαλα που έχουμε στις εκκλησίες, όπου και εκεί είναι θύματα τα παιδιά, να ξέρουμε ότι τις περισσότερες φορές η κακοποίηση ξεκινάει μέσα στο σπίτι. Στηρίζω λοιπόν να συστήσουμε αυτή τη μελέτη. Είπατε ότι πολλές φορές μας λείπουν τα δεδομένα, τα στοιχεία αναλυμένα. Οπότε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την νομοθεσία, όπως είπε και η κυρία Τεριζα Χιμένεθ, πρέπει προηγουμένως να έχουμε τα στοιχεία για να δείξουμε σε όλες τις κυβερνήσεις ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα με συγκριτικά δεδομένα. Έπειτα είπαμε, το σχολείο. Φυσικά όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά στην οικογένεια, οι δάσκαλοι πρέπει να βγάζουν το φίδι από την τρύπα. Αλλά πρέπει να δούμε τι μέσα διαθέτουν ε, τα σχολεία, πώς μπορεί να βοηθήσει το σχολείο και η κοινωνία. Πέρα από το σχολείο όπου οι δάσκαλοι πρέπει να βοηθήσουν ε, και συνήθως δεν επιδέχεται βοήθεια αυτό που έχει συμβεί στο σπίτι, αλλά επιπλέον θα έπρεπε να δούμε μήπω, μια σχολή γονέων κάποτε υπήρχε, στην Ισπανία υπήρχε. Πρέπει να υπάρχουν σχολές κατά κάποιο τρόπο και για τους γονείς μέσα στις δημόσιες δικήσεις, να γίνονται εκστρατείες δηλαδή και για αυτούς, ώστε να μαθαίνουν και εκείνοι. Μια καλή πρακτική για την οδική ασφάλεια. Ήτανε μια εκστρατεία καλών πρακτικών, γιατί μπορεί να υπάρχει νομοθεσία, αλλά δεν τηρείται. Μια εκστρατεία λοιπόν με ευρωπαϊκούς στόχους, ώστε <clears throat> όλοι να ξέρουν ότι κάθε χρόνο θα υπάρξει μέτρηση για να δούμε τι βελτίωση υπάρχει. Αυτό το κάναμε για την οδική ασφάλεια και βοήθησε πολύ. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και εδώ. Τέλος. Πρέπει να ζητήσουμε και περισσότερη συνοχή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που κάνει το ένα χέρι που κόβει δημόσιες επενδύσεις. Να ξέρουμε ότι μετά πού πάνε αυτά τα χρήματα. Από πού μάλλον τα στερούμαστε αυτά τα χρήματα. Να ξέρετε το τι κάνει το άλλο, με δύο λόγια. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Βαλίνα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη, αλλά η ψηφοφορία κράτησε περισσότερο και δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακούσω τις παρεμβάσεις σας, αν το ήθελα πολύ. Θέλω να ρωτήσω γιατί το πιο δύσκολο και το πιο σημαντικό είναι να ξέρουμε την ψυχολογική βία που δύσκολα αποδεικνύεται γιατί στα παιδιά τους κοστίζει πολύ και να την εντοπίσουν και να την εξηγήσουν. Δεν ξέρω, το έχετε λάβει υπόψη σας αυτό το θέμα της ψυχολογικής βίας, πώς αντιμετωπίζετε και πώς εντοπίζετε. Έπειτα στην Ισπανία έχουμε καταστάσεις ουρολιστικές. Διάβαζα για μια δικαστική απόφαση για ένα παιδί που καταδικάστηκε, ένα κορίτσι, ο πατέρας του πέντε χρόνια και όμως επέτρεψαν τις επισκέψεις του πατέρα και μάλιστα χωρίς την παρουσία τρίτου. Ακούω λοιπόν τέτοιες αποφάσεις που δίνεται η κυδαιμονία ε, στον πατέρα παρά το γεγονό ότι υπάρχει κακοποίηση. Γιατί? Γιατί πήγε σε άλλο δήμο να δουλέψει η μητέρα επειδή εκεί βρήκε δουλειά. Και ο δικαστή έτσι αποφασίζει ότι το πατέρα θα κρατήσει το παιδί. Ενώ υπάρχει ενδοοικογενειακή βία. <clears throat> Οπότε και η δικαιοσύνη πρέπει να αλλάξει νοοτροπία και να αντιμετωπίσει διαφορετικά τα παιδιά και τις γυναίκες. Η πατραρχική κοινωνία ξέρουμε τι είναι. Αλλά όταν υπάρχει βία και υπάρχουν ε, άνθρωποι που έχουν ήδη καταδικαστεί, ε, δεν μπορεί να συνεχίσουν να έχουν τέτοια δικαιώματα. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό. Και βέβαια για την κατάρτιση. Γιατί συχνά στη δικαιοσύνη συμβαίνει αυτό και στην Ισπανία έχουμε δικαστικές αποφάσεις που μας εκπλήσουν νομίζουμε ότι βρισκόμαστε σε άλλους αιώνες. σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχουμε 10 λεπτά ακόμα και θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Δύο λεπτά παρακαλώ, γιατί πρέπει να τελειώσουμε στις 12.30 και ακριβώ. Παρακαλώ. Δύο λεπτά. Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι η δικαιοσύνη στην Ισπανία είναι χειρότερη από ό,τι αλλού στην Ευρώπη. Έχουμε βεβαίω περιπτώσει συγκεκριμένε. Εγώ ήθελα να αναφερθώ στη σύγχυση που υπάρχει μεταξύ των δικαιωμάτων των παιδιών, των συστημάτων προστασία επίση, αφετέρου μάλλον, έναντι κρουσμάτων βία μεταξύ των φίλων. Χρειάζεται να έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μα που μπορούμε για να προστατεύσουμε του ανελίκου, αλλά έχουμε και άλλε συμβάσει που είναι άμεσα εφαρμοστέ που, λένε, που προλέπουν άλλα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν μια σύγχυση η οποία οδηγεί πολύ συχνά σε αυτές τις ε, κάπως παράλογες αποφάσεις των δικαστηρίων. Χρειάζεται να γνωρίζουμε το καθεστώς του θύματος και το οποίο μετεγγράφει στην Ισπανία χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας το, την προέλευση, ε, ε, τέλος πάντων τη συγκεκριμένη οικογενειακή προέλευση των γονέων. Καλή η οδηγία του 2012 αλλά με γράφει οδηγία στην Ισπανία χωρίς να συνοδεύεται από μέτρα ε, ειδική ε, ακαθοδήγηση σε περίπτωση ξένων εμπικών. Τώρα τι άλλο να σα πω, υπάρχουν χιλιάδε περιπτώσει. Πριν από δύο μήνε ε, δολοφονήθηκαν δύο κορίτσια στην Καστελιόν αφού είχε γίνει καταγγελία στις υπηρεσίες ε, της κοινωνικής και της υγείας και όπου γνωρίζανε δηλαδή οι υπηρεσίε ότι δεν, δεν υπήρχαν συγκεκριμένε προποθέσει που δεν γινόντουσαν σεβαστέ. Πολύ συχνά δηλαδή παλεύουν οι οικογένειε ή τα μέλη των οικογενειών, όπω μα έδωσε και η κυρία από την Ιταλία, απέναντι στην, στην, στο μέρο τη οικογένεια του πατέρα και αγωνίζονται έναντι προ, προκαταλήψεων και, και, και διοικητικών μέτρων που δυσκολεύουν τη ζωή τους αλλά πρέπει να αναλυθεί αυτή η ευθύνη του γεγονότος ότι μάλιστα πρέπει να αποφύγουμε την επανάληψη τέτοιου είδους ε, ε, συμπεριφορών από πλευρά των παιδιών που έχουν υποστεί τη βία στο μέλλον. Πιστεύω ότι ένα από τα πιο ε, καλά πράγματα τα οποία συνέβησαν σήμερα είναι ότι αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο ζήτημα, μιλάμε για αυτό και με βάση τα όσα είπε η Σουηδέζα Ευρωβουλευτής, ε, οι οργανώσεις θα πρέπει ε, να συνεργαστούν ούτως ώστε να μην επιβάλλουμε τα δικαιώματα των ενηλίκων στα δικαιώματα εις βάρος των δικαιωμάτων των παιδιών. Πιστεύω ότι υπάρχει γνώση όσον αφορά ε, την επιρροή της ενδοοικογενειακής βίας στις δικαστικές αρχές, όμως όχι αρκετή, εξαρτάται από το δικαστή και αυτό λοιπόν δεν είναι αρκετό. Όσον αφορά τώρα την κατάρτιση, Συμπτωματικά την επόμενη εβδομάδα αρχές Δεκέμβρη ε, θα ε, παράσχω ε, εκπαίδευση, ένα σεμινάριο για αυτό το θέμα. Επίσης διδάσκω στο Πανεπιστήμιο φοιτητές νομικής το οποίο επίσης θεωρώ ότι είναι κάτι θετικό, αλλά παρόλα αυτά και άλλα πρέπει να γίνουν. Αυτά, λίγο πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την ε, νομοθεσία, γνωρίζουμε ότι κάποιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν επικυρώσει ακόμα ε, την ε, απαγόρευση της σωματικής τιμωρίας. Δεν έχω εύκαιρη την, τον κατάλογο, όμως αν θέλετε μπορώ να σας, την, να σας στείλω τον κατάλογο αυτών των χωρών. Οπότε ε, ε, όλες οι χώρες θα πρέπει να επικυρώσουν την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και αν υπάρχει δυνατότητα το ίδιο θα πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως επίσης και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών το οποίο δείχνει μεγάλη δέσμευση για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και την καταπολέμηση της βίας με βαστοφύλλο. Ε, η Ρουμανία, ε, έχω εργαστεί εκεί και παρόλο που ε, στα χαρτιά έχει την απαγόρευση της άσκησης σωματικής τιμωρίας, αυτό δεν σημαίνει ότι το εφαρμόζει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα σημαίνει ότι υπάρχει υποχρέωση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. Η έρευνα τώρα θα είναι κάτι το οποίο θα χαρούμε να λάβουμε είναι σημαντικό σε όλα τα δεδομένα και σε όλες τις ε, νομοθεσίες ε, να μην ξεχνούμε τις πιο ευάλωτες ομάδες. Ε, τα εγγόνια μου αναφέρθηκαν πολλές φορές, τώρα το, ε, αναφέρονται εγγόνια. Το αν αυτά υπάρχουν ή όχι, ανήκουν στην οικογένεια όχι, το παιδί είναι παιδί. Ε, κάθε χώρα στην Ευρώπη έχει την υποχρέωση να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν στην περιφέρειά τους. Οι συμβάσεις είναι ξεκάθαρες ότι δεν μπορούν να υπάρχουν διακρίσεις ε, ε, ανάλογα με, τα, με την καταγωγή και την προέλευση των παιδιών. Είναι μια αρχή την οποία θα πρέπει να εφαρμόσουμε στην Ευρώπη και η έρευνα και οι νομοθεσίες θα πρέπει να διασφαλίσουν την πρόσβαση των παιδιών στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Τώρα όσον αφορά την κατανομή των ευρωπαϊκών ε, πόρων ε, σε προγράμματα για την καταπολέμηση της ε, βίας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει, στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο επόμενο ΠΔΠ ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Η προστασία των παιδιών στο τρέχον ΠΔΠ δεν είναι επαρκής και δεν αναφέρεται επαρκώς και ορθά στην προστασία των παιδιών οπότε θα πρέπει αυτή τη φορά να συμπεριληφθεί όπως επίσης και η προστασία από τη βία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πολλά έχουν ήδη υποθεί. Ναι, συγκριτικές μελέτες βεβαίως, συλλογή δεδομένων, ναι, δικτύωση, συντονισμό. Γιατί συχνά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο της Ευρώπης, ε, κάνετε τις ίδιες μελέτες και δεν υπάρχει αρκετή ανταλλαγή πληροφοριών. Οπότε θέλω να ρωτήσω αυτό που είπατε, μιλήσατε για την καλλιέργεια του δικαίου, το δίκαιο ε, του παιδιού, της γυναίκας ε, λοιπά συνδέονται μεταξύ τους, αλλά πρόκειται ακριβώς για μια νοοτροπία δικαίου. είναι ακριβώς είναι που πρέπει να καλλιεργήσουμε. Και εμείς κάνουμε κάτι φιλμάκια για τα παιδιά. Όταν συζητάμε για τη δημοκρατία στα παιδιά, ναι, τι λένε τα παιδιά, ναι, τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε αυτό, σε εκείνο, ε, οι μεγάλοι σε αυτό, εμείς το άλλο. Ε, δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση πρέπει όπου και να βρισκόμαστε να ξέρουμε ότι το δίκαιο μας συνοδεύει, ότι έχουμε δικαιώματα τα οποία δεν είναι υποκειμενικά και πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε και όχι εξ κατέντρα. Φυσικά και στα σχολεία, αλλά παντού η πολιτική νεολαία σε όλα τα στάδια και στην οικογενειακή πολιτική πρέπει να προβλέψει την εκπαίδευση αυτή. Πρέπει να υπάρχει εκδημοκρατισμός του δικαίου και πώς με καινοτομία, με φιλμάκια, με παιχνίδια, με διδακτικό υλικό, ε, το οποίο να είναι διαδραστικό. Και έτσι μπορεί να αλλάξει η νοοτροπία της πρόληψης. Πώς να φτάσουμε στα παιδιά. Δεν θα φτάσουμε με τα βιβλία που θα επιβάλλουμε στο σχολείο. Όχι, με διάφορες εφαρμογές. Τώρα υπάρχουν ψηφιακά. Με καινοτόμα μέσα λοιπόν θα το κάνουμε. Με μέσα το οποίο θα κάνουν το παιδί να ενδιαφερθεί για τα δικαιώματά του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό είναι που πρέπει να φροντίσουμε να διαδοθεί. Γιατί η νομοθεσία φυσικά και είναι πολύ βασική, αλλά δεν γνωρίζει κανείς τι ισχύει και τις έννοιες, δεν τις καταλαβαίνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το θέμα, την οτροπία του δικαίου. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ όλους τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους. Όλοι όσοι είμαστε εδώ και συμμετείχαμε, θεωρήσαμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ακριβώς επειδή είμαστε πολιτικοί, ευρωβουλευτές, να σας ακούσουμε. Η ακρόαση αυτή είναι πολύ σημαντική και ευχαριστούμε και τους επισκέπτες μας από την Ισπανία και την Ιταλία. Σας ευχαριστούμε όλους και όντως πρέπει να συνεργαστούμε για να έχουμε καλά αποτελέσματα και να μπορούμε έτσι να προστατεύουμε τα παιδιά. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. And, uh, next our meeting on the 27 of 27 Νοεμβρίου είναι η επόμενη συνεδρίαση από τις 9 το πρωί, όλη την ημέρα. Ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, και τη Γραμματεία